Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Ξεκινάμε την συνεδρία της Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. First of welcome everybody. Καλώς ήλθατε, καταρχήν, μετά από τις ε, σχολικές διακοπές και ελπίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι να εργαστούμε εποφελώς στο δεύτερο αυτό τμήμα του έτους. Πολλά έχουμε να πράξουμε και είναι υπερπλήρηση η μέρηση διαταξή μας σήμερα και αύριο. Καταρχήν, θέλω να σας ζητήσω, εάν εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη, η οποία σας έχει διανεμηθεί ηλεκτρονικά. Έχετε, προ... έχετε προτάσεις τροποποίησης τη διάταξης, όχι, από ό,τι βλέπω. Η έγκριση λοιπόν τη ημερησίας ε, διάταξης είναι δεδομένη. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Το οποίο είναι η έγκριση των πρακτικών το σχέδιο πρακτικών της 7ης Ιουλίου 2014 και της 23ης Ιουλίου επίσης του ιδίου έτους είναι στα έγγραφα εργασία σας. Εάν, ως συνήθως, δεν εγερθούν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, να θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά αυτά. Έχετε αντιρρήσεις. Παρατηρήσεις για τα πρακτικά της συνεδρίασης 7ης 23ης Ιουλίου. Δεν βλέπω. Ευχαριστώ και πάλι. Θεωρούμε ότι έχουν γίνει δεκτά τα πρακτικά λοιπόν. Τρίτο σημείο της ημερησίας διάταξης είναι η έγκριση του σχεδίου χρονοδιάγραμματος των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ρέτζου για το 2015. Το σχέδιο και πάλι βρίσκεται στο φακελό σας για το 2015 πρέπει να σας αναφέρω ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες για το σχεδιασμό των συνεδριάσεων επιτροπών και αντιπροσωπιών και που είναι υπεύθυνα για την κράτηση αιθουσών και διερμηνέων έχουν κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση την οποία πρέπει να εγκρίνουμε. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις ενδεχομένως για την πρόταση αυτή, για το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, ε, σχόλια για το χρονοδιάγραμμα αυτό που σας έχουμε διανύμει. Όχι. Δεν βλέπω καμία πρόταση, δεν βλέπω καμία αίτηση τροποποίησης. Μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι έχει εγκριθεί και το χρονοδιάγραμμα. Τέταρτο σημείο στην ημέρηση διαταξή μας είναι οι ανακοινώσει της Προέδρου θα μείνετε εμβρόντιτοι, αλλά δεν έχω καμία ανακοίνωση. Μπορούμε να περάσουμε στο πέμπτο σημείο, που είναι η ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Γκρατσάνο δεβιο ο οποίος είναι υφυπουργό και αρμόδιος για τα περιφερειακά θέματα σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας. Όπως ξέρετε, πάντα προσκαλούμε τον αρμόδιο υπουργό ενώπιον της Επιτροπής μας για ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις προτεραιότητες της κατά περίπτωση Προεδρίας του Συμβουλίου. Σήμερα χαιρόμαστε που μπορούμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γκρατσιάνο Δεδίο, από, το, από την ε, Ιταλική Προεδρία η οποία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου. Είναι δυσχερής η εποχή αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχόμαστε στο κύριο Υπουργό και στην Ιταλική Προεδρία κάθε επιτυχία. Ο κύριος Δελρίο είναι ένας από τους πιο ε, εξέχοντες πολιτικούς και συμβούλους του Πρωθυπουργού κυρίου Ρέντσι. Το 2013-2014 ήταν Υπουργός Γενικών Υποθέσεων στην κυβέρνηση του κυρίου Λέτα και έχει περάσει περίπου ε, μία δεκαετία ως ε, δήμαρχος του, της Ω πρόεδρος τη ε, Reggio Emilia. Γνωρίζει λοιπόν πολύ καλά την ε, πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική. Είναι πολύ ενδιαφέρον το βιογραφικό του και εντυπωσιακό και με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε τις απόψεις για την περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω να ακολουθήσουμε την εξή διαδικασία. Θα προσκαλέσω τον κύριο Υπουργό να κάνει μια σύντομη παρουσίαση. 15 περίπου λεπτά σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας στον τομέα φυσικά που είναι αρμόδια η Επιτροπή μας και στη συνέχεια θα έχουμε ε, ερωτήσεις και απαντήσεις σε δύο γύρους ξεκινώντας με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 4.30 για αυτή τη συζήτηση και έχω λοιπόν τη χαρά να δώσω στον κύριο Υπουργό το λόγο. Thank you very ε, ε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε Μιχαήλοβε, αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα του εξαμήνου της Ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την πολιτική συνοχής και για να συζητήσω μαζί σα για τι ερωτήσει, τα θέματα που θεωρείτε πιο σημαντικά. Ο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίω με την Επιτροπή που ασχολείται με την Περιφερειακή Ανάπτυξη είναι τη άμεση αρμοδιότητά μας. Ασχολούμαι δηλαδή με την πολιτική συνοχή και είναι μεγάλη ευκαιρία που έχουμε αυτό ο διάλογος ε, να συζητήσουμε μαζί και η Ιταλική Προεδρία φυσικά θα τον προωθήσει. Θα εστιάσω σε τρία σημεία, καταρχάς πριν μπούμε στο διάλογο. Καταρχά θα αναφερθώ στο πρόγραμμα της Ιταλικής Προεδρία και στο ρόλο τη συνοχή. Θα σα παρουσιάσω κάποιου προβληματισμού για τα βασικά στοιχεία του νομοθετικού πακέτου 2014-2020 και θα κλείσω με τι πρωτοβουλίε που θα προωθήσουμε στα πλαίσια τη πολιτική συνοχή, στα πλαίσια του εξαμήνου τη Προεδρία μα, για να αξιοποιήσουμε κάποιε σημαντικέ καινοτομίε που εμπεριέχονται στα νέα νομοθετικά κείμενα του κανονισμού. Το πρώτο σημείο είναι το πρόγραμμα τη Προεδρία και ο ρόλο τη συνοχή το συνολικό σενάριο στο οποίο, μέσα στο οποίο η Ιταλία ανέλαβε την Προεδρία ε, ρυθμίζεται από την έναρξη ενός νέου πολιτικού κύκλου ε, στη ζωή των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Καταρχάς είχαμε το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές και ανάλογες σημαντικές εξελίξεις ε, συμβαίνουν και στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ιταλική Προεδρία θέλει να βοηθήσει σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, παρά τα πρώτα σημάδια ε, βελτίωσης, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από την Eurostat, που μιλάνε για ανάπτυξη, ε, δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται μέτρα ε, υποστήριξης της ανάπτυξης. Αυτό αφορά όλα τα κράτη-μέλη είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, κυρίως σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής. Ε, πρέπει να σας πω κάποια βασικά στοιχεία. 25 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες είναι άνεργοι και 5 εκατομμύρια από αυτά είναι κάτω από τα 25 χρόνια. Περίπου το 1 τέταρτο της, ε, της, ε, του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κινδυνεύει α, από το φάσμα της φτώχειας και την κοινωνικό αποκλεισμό. Έχουμε και αύξηση 6,5 εκατομμύρια άτομα άνεργοι επιπλέον μεταξύ του 2008 και 2012. Η πρόσφατη οθέτηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκτη έκθεση τη οικονομική και κοινωνική συνοχή και εδαφική συνοχή είναι μια τεράστια και πολύ σημαντική βάση ε, για να προβληματιστούμε και να αναπτυχθούμε. Να σα υπενθυμίσω το στοιχείο τη έκτη έκθεση που μιλάει για το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Μεταξύ του 2008 και του 2013 οι δημόσιε επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 20% σε πραγματικού όρου και αυτή η μείωση θα ήταν ακόμα προφανώ πιο σημαντική αν δεν υπήρχε υποστήριξη από την πολιτική συνοχή. Είναι στοιχεία που δείχνουν ε, σοβαρέ δυσκολίε που πρέπει να υπερκεράσουμε, ε, μια τεράστια κοινωνική αμηχανία ε, και εμφανίζονται ε, με τρόπο ασυμμετρικό στι διάφορε περιοχέ και τα διάφορα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ξέρει πολύ καλά τα ξέρουν πολύ καλά τα μέλη σας. Επαναλαμβάνω κάτι που υποστηρίξαμε ως χώρα στο πρόσφατο φόρουμ, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Συνοχή. Αυτή η Ευρώπη δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη ούτως ώστε να εμφανιστούν ξανά ε, θετικά σημάδια. Η Ιταλική Προεδρία ε, προωθεί τρεις ε, στρατηγικές γραμμές, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση γυπνίαση της Ευρώπης στους πολίτες ε, σε σχέση με την ε, δημοκρατία, τα δικαιώματα και την ε, ελευθερία και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο, σε διεθνές επίπεδο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και στην Επιτροπή σας είναι φυσικά η ανάπτυξη και η απασχόληση. Θέλω να υπενθυμίσω διάφορα στοιχεία που είναι σημαντικά του προγράμματος της Ιταλικής Προεδρίας ακριβώς για αυτά τα θέματα. Καταρχάς, η συνεισφορά που θέλουμε να δώσουμε αφορά την αναθεώρηση και βελτίωση των δεδομένων που σας ανέφερα και τη στρατηγικής Ευρώπη 2020 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμπληρώσει και θα ολοκληρώσει την επόμενη χρονιά. Φυσικά όμως θέλει να ξεκινήσει ο προβληματισμός από τώρα. Προωθούμε ακριβώς γι' αυτό μια ανοιχτή συζήτηση στις διάφορους, στους διάφορους σχηματισμούς του Συμβουλίου για τους τρόπους που θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και αυτός ο προβληματισμός θα γίνει και στα πλαίσια μιας ειδική συνόδου αφιερωμένη στην συνοχή στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου. Θα μιλήσω όμως γι' αυτό αργότερα στην παρέμβασή μου. Ένα άλλο στοιχείο αφορά την ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής διάστασης της ε, Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Εδώ υπάρχει μια πρωτοβουλία δική μας, θα επανέλθω σε αυτήν. Ε, συγκαλέσαμε μια άτυπη υπουργική συνεδρίαση των υπεύθυνων υπουργών για την πολιτική συνοχή που αφορά τη σχέση μεταξύ οικονομικής διακυβέρνησης και πολιτικής συνοχής. Η Ιταλική Προεδρία, στα πλαίσια των μέτρων για την ανάκαμψη, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους υποστήριξης της πραγματικής οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα, του τομέα της βιομηχανίας και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι όλες αυτές οι δράσεις θα πρέπει να δώσουν καρπού στον τομέα της απασχόλησης και κυρίως την απασχόληση των νέων. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχει ήδη προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το σημαντικό τομέα. Η εγγύηση για τους νέους και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι σαφές ότι η πολιτική συνοχή παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μπορεί να βοηθήσει έντονα. Θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή είναι η, πολιτική ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο βασικό μοχλό υποστήριξη ε, για την ανάπτυξη στα πλαίσια τη στρατηγικής Ευρώπη 2020. Είναι εκ των κάνθη για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ε, Έχει πολλά πλεονεκτήματα και σημαντική για τη βιωσιμότητα. Η υποστήριξη τη επιτροπή σα για, το... για την περιφερειακή ανάπτυξη υπήρχε και πιστεύω θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον. Πρέπει να παρέμβουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα για να ενισχύσουμε τις προοπτικές ανάκαμψης. Και αυτό φαίνεται ε, σε κάποιους προβληματισμούς των κοινωτικών θεσμικών οργάνων. Κάθε φορέας θα πρέπει να παίξει το ρόλο του, κάθε θεσμικό όργανο, ή τα κάτι μελη ή κομισιόν, οι πάντες. Και αυτό είπε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου σε σχέση με την στρατηγική ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα πέντε χρόνια, όπου η απασχόληση, η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο επόμενος πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Juncker, το οποίο ευχόμαστε καλή τύχη, θα παρουσιάσει τους πρώτους μήνες ε, μετά την ανάλυση των καθηκόντων του ένα ε, σχέδιο επενδύσεων επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ για τα πρόσφατα τρία χρόνια. Και ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, ο Ντράγκη, ε, μίλησε για την ανάγκη να έχουμε ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Η υποστήριξη της ε, Κεντρικής Τράπεζας είναι πολύ σημαντική. Ξέρουμε ότι δεν υποκαθιστά τα κράτη-μέλη, τα συμπληρώνει για τις απαραίτητε ε, διαθωτικές αλλαγέ. Σε ό,τι αφορά την Ιταλία, να σας πω, δεσμευόμαστε 100% σε... να προωθήσουμε πολύ σημαντικέ μεταρρυθμίσει σημαντικές για την ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020 και την ανταγωνιστικότητα. Παραδείγματο χάρη ε, συνταγματική μεταρρύθμιση, ε, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, δικαιοσύνη, αγορά εργασίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Η πολιτική συνοχή μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο να βοηθήσει την, την Ευρώπη να ξανακερδίσει την ανάκαμψη. είναι σημαντικό ότι το η πλήρη χρησιμοποίηση των διαφορετικών ταμείων ε, είναι σημαντικό για να υλοποιηθεί η, ατζέντα για την, ε, στρατηγική ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το είπε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι η αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα πρέπει να είναι η ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που μας παρέχει η πολιτική συνοχή. Θα ήθελα να φτάσω τώρα στο δεύτερο σημείο της ε, παρέμβασή μου που αφορά τα βασικά στοιχεία του νομοθετικού πακέτου 2014-2020. Ε, Με μια, μετά από μια δύσκολη επραγμάτευση που κράτησε πάνω από δύο χρόνια, το Δεκέμβριο πέρυσι φτάσαμε σε συμφωνία για το νομοθετικό πακέτο για την που αφορά τη συνοχή για την περίοδο 2014-2020. Ευχαριστώ εκ νέου το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για τη δουλειά που κάνανε για αυτό το περίπλοκο ε, και πλήρε θέμα που είναι πολύ σημαντικό για του Ευρωπαίου πολίτε. Χάρη στην ε, ουσιαστική συμμετοχή του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει για την περίοδο 2014-2020 ε, ένα σημαντικό ποσό για τις δημόσιες επενδύσεις, 366 δισεκατομμύρια ευρώ με σημερινές τιμές. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας και την εθνική συγχρηματοδότηση, το ποσό ξεπερνάει 450 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι ένα σημαντικό ποσό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 100% λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα πρέπει να παντρέψουμε μία ε, σφιχτή διαχείριση των ε, δημόσιων οικονομικών και παράλληλα επενδύσεις ε, και μέτρα για την ανάπτυξη. Ε, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2013 για τις ε, τοπικές αρχές ε, και περιφερειακές αρχές ε, και, τις, και τα έξοδα και τα κονδύλια από τα διαφορετικά ταμεία, καθώς και διάφορες αναλύσεις έδειξαν τη σημασία να αποκλείσουμε από τον υπολογισμό το σχέδιο σταθερότητας και ανάπτυξης ή μάλλον από το σχέδιο σταθερότητας και ανάπτυξης την εθνική συγχρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής. πρέπει να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ε, και αυτό δεν είναι αντίθετο από τις ε, δημοσιονομικές επιταγές. Πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας την οικονομική διακυβέρνηση και το στενό σύνδεσμο με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, στην μακροοικονομική ερεσιμότητα Και αυτό ε, θα μπορούσε να συζητηθεί στα πλαίσια της, υπουργικής, της άτυπης υπουργικής διάσκεψης 10 Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το βασικό στοιχείο της ε, συνεδρίασης είναι να δούμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής συνοχής και οικονομικής διακυβέρνησης. Θα ακούσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και την συνεισφορά της Προέδρου Μιχαήλοβα. Ε, υπενθύμησα αυτά τα ποσοτικά στοιχεία του νομοθετικού πακέτου της συνοχής για το 2014-2020 γιατί είναι πολύ σημαντικό, σημαντικά στοιχεία και αφορούν και την κοινή μας δουλειά. Θέλω να σας πω ότι πέρα από τη χρηματοδότηση όμως Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι η ποσότητα και η αποτελεσματικότητα τη χρήση αυτών των ποσών. Και ακριβώ το νομοθετικό πακέτο αυτό τονίζεται με πολύ έντονο τρόπο. Έχουμε κοινό καθήκον να διοχετεύσουμε τα κονδύλια τη πολιτική συνοχή με τρόπο ούτω ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Να σα ε, υπενθυμίσω ότι για την ποιότητα ε, θα πρέπει να προσανατολιστούμε στα αποτελέσματα, που είναι το βασικό στοιχείο τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποστήριξαν στη διαπραγμάτευση. Και τώρα είναι τμήμα του νομοθετικού πακέτου. Η λογική των παρεμβάσεων θέτει στο κέντρο τι ε, θετικέ αλλαγέ για του πολίτε και τι επιχειρήσει μετά από τι επενδύσεις. Θα πρέπει δηλαδή να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα Όποιος και είναι ο θεματικός στόχος της επένδυσης, ε, έρευνα, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κτλ. Οι κανόνες ε, για την τρέχουσα περίοδο απαιτούν να έχουμε συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα στοιχεία προόδου με τα κονδύλια αυτά. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και θα πρέπει να ε, είναι θετικά τα αποτελέσματα και για τους δικαιούχους αλλά και για τους πληρωτές. Επίσης, κάποια άλλα στοιχεία βασικά για την περίοδο 2014-2020. Η σχέση ε, μεταξύ της ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, η, στρατηγική, Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 και οι συστάσεις αναχώρα. Η εισαγωγή της εξάντε αιρεσιμότητας, η θεματική συγκέντρωση Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Και η μεγαλύτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην εταιρική σχέση, ε, όλα αυτά θα συντελέσουν την επιτυχία. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ, θα ήθελα να μιλήσω ξανά για την ευγνωμοσύνη που έχω για τον συμβασμό που επετέχθη μετά από μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση για αυτό το σύνολο ε, καινοτόμων κανόνων. Πολλά από τα στοιχεία που ανέφερα για, αυτές, για τους κανονισμούς, παραδείγματο χάρη ο κώδικας διοντολογίας ε, για την εταιρική σχέση. Οι πολλές ε, αλλαγές για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα προκύπτουν από την διαπραγματευτική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην φάση ενεργοποίησης του και προγραμματισμού της περίοδου 2020, όπου θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει ε, μαζί να βοηθήσουν τόσο ώστε να γίνουν αποτελεσματικές αυτές οι αλλαγές ούτως ώστε μετά από λίγα χρόνια να έχουμε τις πρώτες απτές βελτιώσεις στα διάφορα θεματικούς, διάφορους θεματικούς τομείς όπου συγκεντρώνονται οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής. Θέλω να μιλήσω τώρα για κάποιους πρωτοβουλίες του εξαμήνου. Η Ιταλική Προεδρία προσπάθησε να μιλήσει για μια νέα ε, συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις ευκαιρίες και για να είναι πιο αποτελεσματική η συνεισφορά στην πολιτική ε, συνοχής. Θα ήθελα να υπενθυμίσω καταρχάς ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την θέση σε ισχύ των κατεξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται στον κανονισμό και που η Κομισιόν θα υιοθετήσει κατά τη διάρκεια της ε, του εξαμήνου μας ό,τι αφορά την ε, εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα και η θα βασιστούμε στη θαυμάσια δουλειά που έκανε η Ελληνική Προεδρία και τις διαδικασίες που ξεκίνησε. Η πιο σημαντική πρωτοβουλία όμως σε πολιτικό επίπεδο αφορά την προώθηση ενός ε, πολιτικού διαρθωμένου διαλόγου στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Όπως ξέρετε η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα είναι, χαρακτηρίζεται από το ότι η πολιτική συνοχής, που όπως σας είπα και προηγουμένως είναι η πολιτική ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι περίπου το 1 τρίτο του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν διαθέτει στα πλαίσια του Συμβουλίου ε, μία πραγματική έδρα ε, πολιτική και τακτική συζήτηση. Η εντύπωση αυτή προκύπτει και μέσω από τις πρωτοβουλίες ελληνικής προεδρίας ε, με την υποστήριξη του Επιτρόπου Χάν. Προσπαθούμε δηλαδή στο κέντρο τη πολιτική συζήτηση και στι εργασίε του Συμβουλίου να θέσουμε το θέμα των πολιτικών συνοχή ούτως ώστε να υπάρχει μια συνείδηση ε, για τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. Θα πρέπει λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο να μπει στο κέντρο το θέμα των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής σε σχέση με, τις, ε, με τους στόχους της στρατηγικής 2020. Πέρα από την άτυπη υπουργική ε, συνεδρίαση που συνήθως γίνεται, μαζί με τις πρωτοβουλίες που είχε ξεκινήσει η Πολωνική Προεδρία του 2011, έχουμε προ προβλέψει ε, στις 19 Νοεμβρίου μία ειδική σύνοδο για την πολιτική συνοχή στα πλαίσια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, γιατί ακριβώς δίδουμε μεγάλη σημασία στην ε, συνοχή και στη συνεισφορά της στην ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω αυτό και για σας. Και θέλω να σας τονίσω ότι αυτός είναι ένας τρόπος για μας για να αναγνωρίσουμε περαιτέρω τη σημασία των καινοτομιών που συμπεριλαμβάνονται στα νέα, στους νέους κανονισμούς και να τα αξιοποιήσουμε πλήρως διάφορες νέες ε, διατάξεις του πακέτου, νομοθετικού πακέτου 2014-2020 αναφέρονται σε έναν ε, ενισχυμένο πολιτικό διάλογο μεταξύ των θεσμικών και κοινωνικών οργάνων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο, με τη συνεισφορά τη Επιτροπή των Περιφερειών και τη ΕΟΚΕ. Αυτό ο διάλογο θα πρέπει να είναι ε, μια νέα όθηση, μια νέα ορμή, επαλήθευση, προβληματισμό, για να δούμε το πώ θα υιοθετήσουμε τι αποφάσει για την ενεργοποίηση και εφαρμογή των επενδύσεων. Όλα αυτά τα στοιχεία ε, τα, συζητήσαμε διαπραγματεύοντα, όταν διαπραγματευτήκαμε το πακέτο 2014-2020. Ε, γύρω από την αρχή ε, ξοδεύουμε καλύτερα, better spending, ε, σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η ενεργοποίηση του προγραμματισμού θα συνοδευτεί λοιπόν από διάφορες διατάξεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, διάφορες εκθέσεις κτλ οι νέοι κανόνες για την μακροοικονομική ερεσιμότητα ε, μιλούν ε, ρητά για το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις αποφάσεις που θα πρέπει να υιοθετεί το Συμβούλιο μετά από προτάσεις της Επιτροπής. Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία, τα νομοθετικά, θα πρέπει να τα παρακολουθεί η Προεδρία για να εξασφαλίσει σε αυτή τη μεταβατική περίοδο στη ζωή των, ε, τη θεσμική μας μια συνέχεια θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο, ούτω ώστε να καταστήσουμε σαφή τη χρησιμότητα της πολιτικής συνοχής. Στην έκτη έκθεση για τη συνοχή έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση ε, και να επικεντρωθούμε ε, στον προγραμματισμό και και να επικεντρωθούμε και στον προγραμματισμό, αλλά και σε διάφορες ε, σκέψεις, σε διάφορους προβληματισμούς. Ε, θέλουμε λοιπόν ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων να συνεισφέρουμε ε, στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 με τρόπο ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη την πολιτική συνοχής και το σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη, τη συνοχή κτλ. Είμαι έτοιμος να συζητήσω μαζί σας για αυτά τα θέματα. Thank Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση αυτή. Νομίζω ότι έχουμε πλέον αρκετές πληροφορίες που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης που θα επακολουθήσει. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στους συντονιστές. Ο κ. Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ πολύ θα μπορούσαμε να έχουμε δύο γύρους ε, ώστε να ακουστούν ως το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές. Θα είμαι σύντομος. Ε, θα σας ευχαριστήσω καταρχάς για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για το έργο που έχετε επιτελέσει. Θα είχα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σύντομε. Πρώτον, αυτή την άτυπη συνάντηση των Υπουργών για την Περιφερειακή Πολιτική που αναφέρατε, αν γίνει, μην δείτε μόνο προς τα εμπρός αλλά και προς τα πίσω. Με την εκτή έκθεση για τη συνοχή παίρνουμε πολλά στοιχεία, ε, αλλά κυρίως για τις πληρωμές πρέπει να δούμε. Διότι άκουσα μεταξύ άλλων σε αυτό το, για αυτό το έκτο φόρουμ για τη συνοχή, ότι όλοι μιλάνε για το μέλλον και για το απότερο μέλλον. Είπατε αυτά τα 300 εκατομμύρια, το φρέσκο χρήμα που πρέπει να βρει ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δημιουργήσει, αλλά ας δούμε τις επιδόσεις μας, ας δούμε τι γίνεται με τις πληρωμές. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση στην Ιταλία. Σε πολλές χώρες ακούω ότι υπάρχουν λογαριασμοί οι οποίοι μετατίθενται για το 2015 Υπάρχει όλο και πιο διεξοδικός έλεγχος των προγραμμάτων και λίγα πράγματα γίνονται για να περάσουν τα πράγματα στο επόμενο έτος και όλοι είναι απογοητευμένοι για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και είναι κάτι που γνωρίζει, θα γνωρίσει έκρηξη ε, με τις πληρωμές μέσα στον επόμενο χρόνο. Έχουμε διαφορά μεγάλη μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Πώς θα καλύψουν αυτό το κενό, πώς θα μας εμπιστευτεί ο κόσμος, οι επιχειρήσει, οι δημόσιες αρχές, πώς θα καταβάλουν οι δημόσιες αρχές το δικό τους μερίδιο σε συγχρηματοδότηση αν δεν πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας παρακαλώ βάλτε το αυτό το θέμα στην μεσαία διάταξη αυτή της άτυπης συνάντηση. Επίσης είπατε ότι θέλετε να έχετε μια ανοιχτή σχέση, δέσμευση με, τις, με τους οργανισμούς της Ένωσης γενικώς. Μήπω η ευρύτερη συμμετοχή τη επιτροπή Ρέγγι με την πρόεδρό μα αλλά και άλλοι. Θα ήταν κάτι καλό. Επίση, για τι πρωτοβουλίε που αναφέρατε, μιλήσατε για τι δύο συναντήσει τη άτυπες των Υπουργών. Σημαντικό είναι και αυτό, αλλά ε, να έχετε υπόψη σε αυτό που σα είπα για τις πληρωμές και προσθέστε το παρακαλώ στην ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν ε, κονδύλια, δεν θα ξεκινήσουν προγράμματα. Έχουμε και την οδηγία για τι καθυστερούμενε πληρωμέ πρέπει να πληρώσουμε σε 30 μέρες μέσα. Για τους άλλους ισχύει αυτός ο κανόνας, δεν ισχύει για μας. Νομίζω αυτό είναι σημαντικό για το Συμβούλιο. Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Φανή Στελρόη. Κύριος Βον. Ή όχι. Το ελέγχω για να σιγουρευτώ αν πάρω την ε, έγκριση της συντονίστριας. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσίαση. Το πρώτο σημείο έχει σχέση και με αυτό που είπε ο κύριος Φανής δηλαδή το θέμα που έθεσε και αυτός για τον προϋπολογισμό. Με βάση αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2013 είχαμε υστέρηση πληρωμών στο έψος των 23 δις και μας λέει η Κομισιόν ότι στο τέλος του 2014 θα εξακολουθήσει να υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών, 18 δις ευρώ. Και αυτό δυνητικά θα προκαλέσει προβλήματα στους δικαιούχους. Τοπικές αρχές, περιφέρειες, πανεπιστήμια, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, επιχειρήσεις, όλοι αυτοί οι φορείς ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω καθυστέρησης πληρωμών. Εσείς λοιπόν τους επόμενους μήνες πιστεύω ότι έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να εκδεδερματίσετε ώστε να περάσει αυτό το μήνυμα στα άλλα κράτη-μέλη. Πολλά κράτη-μέλη δέχονται αυτή τη θέση αλλά ε, ορισμένα δεν τη δέχονται από ό,τι γνωρίζουμε. Άρα έχετε ένα σημαντικό ρόλο. Πρέπει να πείσετε τα κράτη-μέλη ότι υπάρχει πρόβλημα με τι πληρωμέ. Και αν δεν κάνουν κάτι τα κράτη-μέλη για να επιληθεί αυτό το ζήτημα, οι ΜΚΟ, τοπικέ αρχέ, περιφέρειες, επιχειρήσει, ε, θα έρθουν να παραπονεθούν στι χώρε λόγω των καθυστερούμενων πληρωμών. Άρα, όπω και ο κ. Φανή Τελόρη, σας ερωτώ, ω Προεδρεύον του Συμβουλίου για του προσεχεί μήνε, πώ θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα, πώ θα πείσετε τα άλλα κρατημέλη να αντιμετωπίσουν αυτέ τι καθυστερήσει πληρωμέ. Δεύτερον, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, να μιλήσατε και για, το, ε, για την εγγύηση για την νεολαία. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή καταρτίζουν ε, τα κράτη-μέλη τα σχέδια υλοποίησης. Δεν έχουν ξεκινήσει όμως όλα τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν κάποια κράτη που ξέρουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια της εγγύησης για την νεολαία, αλλά θα τοποθετήσουν τα κονδύλια αυτά σε προγράμματα που ήδη λειτουργούν υπό τη δική τους αιγίδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Ένα λέει κάνει το ένα κράτος, τελείως αντίθετα λέει και πράττει το επόμενο. Πρέπει λοιπόν αυτού του μήνε που θα έχετε την Προεδρία να φροντίσετε να υπάρχει συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ε, το, ε, του Ταμείου Συνοχή. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό ο συντονισμό. Έχετε ρόλο και σα ερωτώ και εδώ τι θα κάνετε για να υπάρξει συντονισμό, να αναλαμβάνουν τα κρατημέλη συντονισμένη δράση και να αξιοποιηθούν τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Πρόεδρος. I didn't spell. I'm sorry for, for the spelling. Λούερ ή κάπως έτσι σας λένε, με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να σας προφέρω σωστά το όνομα. So you, Mr. Jakovčić. Dobar dan i poštovanje Γιάκοφτιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω η Ιταλική Προεδρία να αφιερώσει κάποια προσοχή και στη Μεσόγειο. Εγώ είμαι από την Κροατία, γείτονα δηλαδή. Μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα με την Ιταλία, γι' αυτό θα με ενδιέφερε να ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία στην Αδριατική. Έχουμε τη στρατηγική Αδριατική Ιωνίου. Πώς θα εξελιχθεί η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Και πώς θα συνεργαστείτε και με άλλους ε, επιτρόπους, τον κύριο Χάντη, την κυρία Κρέτου, που θα αναλάβει την περιφερειακή ανάπτυξη ο κύριο Χάν ξέρουμε ότι είναι αρμόδιο για τα θέματα τη διεύθυνση. Ελπίζουμε λοιπόν η Ιταλία να έχει μια σαφή στρατηγική για το θέμα αυτό. Διότι έχουμε τη θάλασσα, έχουμε και την νεολική ενέργεια. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Και έρχομαι σε κάτι πιο γενικό. Είμαι νέος βουλευτής πρώτη θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ήμουν όμως ε, στην κλειστική εξουσία ε, στην Κροατία 20 χρόνια περίπου και με εκπλήσει η πολύ μικρή θέση που βλέπω να έχει ο τουρισμός ε, στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να, να μου πείτε εσείς στο Ιταλικό Κοινοβούλιο που ξέρουμε πόσο σημασία έχει ο τουρισμός για την Ιταλία. Πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι μέσω των πολιτικών συνοχής και εν γέννη με την πολιτική που αποσκοπεί στη βελτίωση της οικονομίας, πιστεύω ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει ο τουρισμός, κυρίως να βοηθήσει τους νέους και αυτούς κυρίως που δεν μπόρεσαν να αποφεληθούν να εκπαίδευσης κατάλληλης, γιατί ξέρουμε ότι τα τουριστικά επαγγέλματα ε, δεν τα σπουδάζει πολύ ε, κόσμος πολύ καλά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον αντιπρόεδρο. Ο Μάρτζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, αναφερθήκατε στην πολιτική σημασία που επέχει η περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές ότι η Επιτροπή μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτή τη διάσταση της ενωσιακής πολιτικής. Και προσπαθούμε να δώσουμε μια σημαντική συμβολή, όπως το πράξαμε και στη διαπραγμάτευση για τα διάφορα ταμεία. Από τη δική σας πλευρά πρέπει να τονίσω ότι έχετε ενώπιόν σας μια επιτροπή που απαρτίζεται από φίλους της περιφερειακής πολιτικής. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον της περιφερειακής πολιτικής. Αλλά, σύμφωνα μαζί σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταδείξουμε το ότι η περιφερειακή πολιτική είναι αποτελεσματική. Ότι τα ταμεία πιάνουν τόπο. Ότι υπάρχει απαραίτητη διαφάνεια στην εφαρμογή των περιφερειακών πόρων και ότι υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι οι οποίοι απαιτούνται για μια πολιτική αυτού του είδους, γιατί έχουμε πολλές φορές επικρίσεις, κυρίως άδικες επικρίσεις, οι οποίες κατευθύνονται κατά της περιφερειακής πολιτικής. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να θέσουμε και το ερώτημα του τι θα γίνει με τα 23 εκατομμύρια ευρώ χρέους στον προϋπολογισμό ποσών δηλαδή τα οποία δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και τις ε, συναφείς ανησυχίες που υπάρχουν για τις πιστώσεις πληρωμών. Προς το παρόν, με διάφορα τεχνάσματα και ακροβασίες μπορούμε να καλύπτουμε τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν, αλλά σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να υπάρξει ένας πιο συνεκτικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και αν θα προκύψουν σοβαρές συνέπειες για τις περιφέρειες της Ευρώπης και τι προβλέψει συγκεκριμένα να κάνει η Ιταλική Προεδρία για το θέμα αυτό. Ένα τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω αφορά την ε, σύνδεση μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών αφενός και της οικονομικής διακυβέρνησης από την άλλη πλευρά. Η λεγόμενη δηλαδή μακροοικονομική ερασιμότητα. Το ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω είναι ποιες είναι οι θέσεις στο εσωτερικό του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για το θέμα αυτό της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Υπάρχει ομοφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί αυτή η σύνδεση με την οικονομική διακυβέρνηση στην περιφερειακή πολιτική ή υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Τέλος, επανέρχομαι στην πρόταση η οποία έγινε από τον κύριο Φανίστ Λερόι να συμμετάσχει η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διάφορες σημαντικές χρονικές ε, στιγμές που ανέφερε, αναφέρατε από την Προεδρία σας, δηλαδή τα ραντεβού αυτά σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Κυρία Βάνα, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να συνεχίσω με αυτά που είπε ο, προ... ο προλαλής σας για τις πληρωμές οι οποίες ακόμα εκκρεμούν και το τι θα γίνει με το έλλειμμα αυτό το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο για την ευρωπαϊκή πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο και που κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνη έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησατε για ένα πρόγραμμα επενδύσεων 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει αναφερθεί και από τον πρόεδρο Γιούνκερ και από την προτινόμενο, το προτινόμενο επίτροπο. Το ερώτημά μου είναι, μέσα στο πρόγραμμα αυτό επενδύσεων που έχει προταθεί, σε ποιο βαθμό θα υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, η αηφόρος ανάπτυξη που έχουμε υποστηρίξει πάρα πολλές φορές. Και εσείς το έχετε αναφέρει το θέμα αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πόσο μεγάλη έμφαση θα δοθεί στις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της αηφόρου λειτουργίας των επιχειρήσεων και φυσικά μας ενδιαφέρει και το θέμα της απασχόλησης, πώς θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την ανεργία των νέων και ένα τρίτο σημαντικό σημείο το οποίο αναφέρατε είναι οι δημόσιες επενδύσεις. Και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στις δημόσιες υπηρεσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο σε επίπεδο περιφερειών και σε πόλεων. Ποιε είναι λοιπόν οι προθέσεις σας σε σχέση με τις ε, επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την παροχή κέριων δημοσίων υπηρεσιών. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Κύριε Νταμάτο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Νομίζω οι περισσότερες ερωτήσεις έχουν εστιάσει στα ίδια θέματα που έχουν να κάνουν και με το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας και με τη βιωσιμότητα των μελλοντικών επενδύσεων στις βιομηχανίες. Μας ενδιαφέρει να έχουμε μια πιο συνεκτική οικονομική δραστηριότητα σε κέριου τομεί όπω είναι παραγωγικά και ο τουρισμό, που είπε ο Κροάτης συνάδελφος. Επιπλέον θέλω να επιστήσω την προσοχή σα σε ένα ουσιαστικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το Σύμφωνο σταθερότητα, που είναι η ανάγκη διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Αυτέ οι μεταρρυθμίσει πρέπει να γίνουν προ το καλό των πολιτών μα και αυτό αφορά ιδιαίτερα τη δική μα μας χώρα την Ιταλία. Ευχαριστώ. Έχουμε κλείσει τον πρώτο γύρο λοιπόν των ε, ερωτήσεων και έχετε εσείς το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θέλω πρώτα απ' όλα να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Είναι από τα πιο σημαντικά θέματα αυτό για την τελική αποτελεσματικότητα των πολιτικών συνοχής. Φυσικά δεν έχει κανένα νόημα οποιαδήποτε δέσμευση αν δεν έχουμε προβλέψει και τις κατάλληλες πληρωμές στον προϋπολογισμό, τις δεσμεύσεις πληρωμών. Η δέσμευσή μας λοιπόν είναι απόλυτη σε αυτό το σημείο. Ξέρουμε ότι είναι ένα σημείο κλειδί για να υπερασπιστούμε τα ταμεία συνοχής. Και όλες οι διαπραγματεύσεις που θα κάνουμε με την Επιτροπή, είναι ε, σε, αυτή την, σε αυτόν τον αγώνα σημαντικό η δική σας ε, συνεισφορά, η δική σας βοήθεια για να διατηρήσουμε αυτά τα κονδύλια. Ξέρετε πολύ καλά ότι έγιναν πολύ σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Υπάρχουν δυσκολίες. Αυτές οι περικοπές αφορούν μόνο μερικώς, ευτυχώς, τα κεφάλαια που αφορούν την πολιτική συνοχή, αλλά θεωρούμε ότι το θέμα των πληρωμών είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που θα πρέπει να απασχολήσουν την άτυπη Υπουργική Σύνοδο των Υπουργών Συνοχής και θα πρέπει να συζητηθεί πάρα αυτά και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 19 Νοεμβρίου. Γιατί οι πολιτικές συνοχής γενικά επηρεάζουν όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα μαζί με άλλα σημαντικά θέματα σε αυτό το σημείο λοιπόν υπάρχει απόλυτη δέσμευση της Ιταλικής Προεδρίας. Σας το εγγυώμαι. Το έχουμε απόλυτα στο μυαλό μας αυτό το θέμα. Έπειτα, μιλήσατε για το θέμα μιας ασυμμετρίας, αν κατάλαβα καλά, όπως είπε ο κύριος Βόγκαν. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα για την απασχόληση ας πούμε των νέων. Νομίζω ότι ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ε, αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δίνει πολλές ελπίδες. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ιταλία είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι για το θέμα της ανεργία των, των νέων. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα εμείς, πολύ ψηλά ποσοστά. Το πρόβλημα που υπάρχει και το υπογραμμίζουμε και θα το τονίσουμε και στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εργασία και Ανάπτυξη και Απασχόληση είναι ότι συχνά υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα κατακαιρματισμένα που τρέχουν παράλληλα και αυτό το, αυτή η εγγύηση των νέων είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί σωστά. Το θέμα του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό των κρατών μελών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κύριε Φανίστελ Ρόι, σας διαβεβαιώ ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τιμήσουμε τους χρόνους πληρωμής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για τις επιχειρήσεις μας, για τα πανεπιστήμια μας, για τα ζωντανά σώματα της κοινωνίας μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για τις αγκαίρες πληρωμές, για την καταβολή των πληρωμών εγκαίρως. Κάποιος άλλο μίλησε για το που έχει φτάσει η στρατηγική για την Αδριατική. Ο βουλευτής από την Κροατία. Έχουμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια για την στρατηγική για την Αδριατική και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε γιατί εμείς θα δώσουμε τεράστια προσοχή και σημασία. Είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι, προφανώς. Είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία εστιάζουμε. Μιλάμε και για την... Ασχολούμαστε πάρα πολύ έντονα και με την μπλε οικονομία, την, τον τουρισμό, την οικονομία της θάλασσας γενικά. Και θέλουμε να, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου να συμπεριληφθεί και το θέμα της Αδριατικής. Αυτά τα συμπεράσματα λοιπόν, εν συνεχεία, θα οδηγήσουν στην εφαρμογή της στρατηγικής και στο συντονισμό για τη στρατηγική. Φυσικά ο τουρισμός είναι ένα από τα στοιχεία και σε κάποια κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, αλλά και άλλα κράτη-μέλη, Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, πολύ σημαντική αυτή η στρατηγική και για την απασχόληση. Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική για την Αδριατική, αλλά και άλλες στρατηγικές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν τον τομέα του τουρισμού. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής σας μίλησε για τους θειασότες και τους πολέμιους της ε, πολιτικής συνοχής. Ε, υπάρχουν στα θεσμικά μας όργανα. Προφανώς, συμφωνώ. Το βασικό πράγμα που θα, σοπάς, κάνει να σοπάσουν οι πολέμοι της ε, πολιτικής συνοχής είναι να παίξει πραγματικά το ρόλο της, να γίνει ένα στρατηγικός ε, προγραμματισμός κατάλληλος για κάθε επικράτεια που θα δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη. Να ξοδευτούν σωστά τα κονδύλια, να προωθήσουμε ε, βιώσιμη ανάπτυξη και σταθερή απασχόληση. Όλοι δεσμευόμαστε, όλοι όσοι πιστεύουμε, όπως και η Ιταλική Προεδρία, πιστεύουμε σε αυτή την πολιτική συνοχή. Και πιστεύουμε ότι οι κεντρικές πολιτικές και οι πολιτικές, οι περιφερειακές πρέπει να πάνε χέρι-χέρι. Είναι σημαντικό για να αναπτυχθεί αρμονικά η Ευρώπη. Αλλά και κάθε χώρα. Το θέμα της διαφάνειας στη χρήση των κονδυλίων των, ταμείων, το θέμα της, του απολογισμού και της λογοδοσίας τη χρήση των κονδυλίων από τα ταμεία. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό. Μια τελευταία ερώτηση για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Υπάρχουν εδώ διάφορες θέσεις, προφανώς, το ξέρετε. Η ισορροπία που επετεύχθη ενός μη αυτόματου μηχανισμού. Ε, να μην αρχίσει να τρέχει αυτόματα δηλαδή, αλλά θα πρέπει να συζητάμε τις συνθήκες ε, της κάθε χώρας. Αυτός είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός για ένα κανόνα που σε πολλά κράτη δημιούργησε πολλές αμφιβολίες που θεωρώ και θεμητές. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη βέβαια. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν θυμάμαι το όνομα της Γερμανίδας βουλευτού που έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Είναι πολύ ε, εξειδικευμένο. Και εμένα με ενδιαφέρει τι θα γίνει με αυτά τα 300 δισεκατομμύρια. Και από αυτά η ποσόστοση για την απασχόληση, ποια θα είναι η ποσόστοση για την ε, βιωσιμότητα. Δεν ξέρω δηλαδή από αυτά τα 300 δις, ας πούμε, πού θα πάει τι. Αυτό δεν το ξέρω. Ίσως θα πρέπει να ρωτήσουμε τον πρόεδρο Γιούνκερ. Βεβαίως, εμείς θέλουμε να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό. Κύριε Μάτο, οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις και η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας για αυτό το, κεφάλαιο των πολιτικών συνοχής. Αυτό ήταν το θέμα του. Τι γίνεται με αυτό. Η άποψη ότι οι πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη είναι το μοναδικό μεγάλο κεφάλαιο που χρειαζόμαστε. Όπως είπα και εγώ στην παρέμβασή μου, νομίζω ότι αυτό συνάδει με στρατηγικές ανάκαμψης της οικονομίας, ε, με στρατηγικές ανάπτυξης και θα πρέπει να δούμε το, τα ποσοστά συγχρηματοδότηση που αποκλείονται από το σύμφωνο σταθερότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω ότι είναι λογικό και πιστεύω ότι μια και πρόκειται για επενδύσεις που τις, έχουμε, τις έχουν ε, συζητήσει οι χώρες και με την Ευρώπη και τις έχει εγκρίνει το ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως δεν τις κάνουν μόνες τους οι χώρες. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει αυτή η εξαίρεση. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν εκ νέου ένας προβληματισμός με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με όλες τις ασφαλιστικές δικλείδεις. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό, ούτω ώστε να γίνεται αυτό παράλληλα με μια προσπάθεια ε, διευκόλυνσης των δημοσίων επενδύσεων ε, για την ανάπτυξη των χωρών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντελρίο. Αγαπητοί συνάδελφοι, για τον επόμενο γύρο έχουμε κάτι παραπάνω από μισή ώρα. Και έχω ήδη αρκετούς συναδέλφους που είναι γραμμένοι στον κατάλογο των ομιλητών. Κυρία Πρέσο. Έχετε το λόγο κυρία Πρέσο. Ε, Ευχαριστώ και σύντομα. Ο Υφυπουργός Δελρίο Μίλησε για την σημαντική πτώση των επενδύσεων. 20% είναι δραματική αυτή η μείωση στην Ευρώπη. Είναι ένας ευρωπαϊκός μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποια τμήματα της Ευρώπης έχουμε πάνω από 20% μείωση των επενδύσεων. Ανάλογα δεδομένα, αντίστοιχα δεδομένα για τις δαπάνες θα μας ε, σκιαγραφούσαν μια διαφορετική πραγματικότητα. Παρά την ανάγκη που έχουμε με βάση τη στρατηγική Ευρώπη 2020 ε, και παρά την, τις πολιτικές συνοχής, ε, πιστεύω ότι δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να βοηθήσουμε την ανάπτυξη, να βοηθήσουμε την απασχόληση αρκετά. Νομίζω ότι αυτό το πολιτικό θέμα, το το πολύ ουσιαστικό είναι καθήκον της Ιταλικής Προεδρίας να το θέσει. Συνδέεται φυσικά με τα 300 δισεκατομμύρια που λέγαμε πριν, που θα πρέπει να είναι επιπλέον και όχι τα μόνα. Έτσι. Και επιπλέον να επιταχυνθεί και να ενεργοποιηθεί περισσότερο η πολιτική συνοχή μαζί με ένα νέο τύπου προγραμματισμό. Καθώς και νέα μέτρα που θα επιτρέψουν στα κράτη τα οποία είναι καλοί μαθητές ε, σε επίπεδο δαπανών, να δώσουν μεγαλύτερη σημασία, σημασία ε, σε σωστές, σε κατάλληλες επενδύσεις. Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, ήρθα λιγάκι καθώς, ε, καθυστερημένα και δεν έχω ακούσει το σύνολο των ε, παρατηρήσεών σας καταρχήν. Είχα καθυστέρηση στην πτήση μου, ήρθα μία ώρα καθυστερημένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας ζητώ συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει, εάν ρωτήσω κάτι που έχετε ήδη πει, μην ε, με ψέγετε, απλώς δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Είναι το θέμα των πληρωμών οι οποίες ακόμα εκκρεμούν, που ήθελα να αναφέρω, δεν είναι καινούριο πρόβλημα. Είναι χρήματα τα οποία είναι κονδύλια τα οποία αναβάλλεται κάθε φορά η καταβολή τους και θα ήθελα εδώ να θέσω ένα ερώτημα. Έχετε εσείς η Ιταλική Προεδρία κάποια συγκεκριμένα σχέδια, κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εγώ βλέπω ότι είναι πραγματικά παράλογο να μιλάμε από τη μια μεριά για προγράμματα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Είναι σε πολλά κράτη-μέλη το πρόβλημα αυτό ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία εκτελέστηκαν, αλλά στη συνέχεια δεν μπορούν να καταβληθούν οι απαραίτητε πληρωμές. Αυτό δεν βοηθάει τον πληθυσμό να έχει μια ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε τους ε, παροτρύνει να συνεχίσουν να επενδύουν σε παρόμοια σχέδια. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν έχετε κάποια συγκεκριμένη απάντηση στο, στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και αν θα υπάρξει κάποια πρόεδρος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Ελπίζω λοιπόν ότι από την Ιταλική Προεδρία θα προέλθει κάποια πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερον, έχω ένα ερώτημα ακόμα. Είναι σχετικά περιορισμένες οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί. Έχετε και εδώ κάποια πρωτοβουλία με την οποία εσείς θα μπορέσετε, εφόσον το επιθυμείτε φυσικά, να πιέσετε τα κράτη-μέλη και να τα βοηθήσετε ώστε να έχουν την απαραίτητη αρρωγή για να δράσουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, ενώ κάποια άλλα έχουν λιγότερη εμπειρία, αλλά είναι φυσικά προς το συμφέρον των ίδιων των κατών μελών, το ταχύτερο δυνατό να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά τα προγράμματα. Και επίσης, στη συνέχεια αυτού που ανέφερα για τα προγράμματα τα λειτουργικά που δεν έχουν εγκριθεί, τουλάχιστον δεν έχουν εγκριθεί όλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια καθυστέρηση και αυτό δεν βοηθάει καθόλου, ιδίω για τις πρωτοβουλίε που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Έχετε κάποια ιδέα για το αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποιος μεταβατικός κανονισμός ώστε να μην καθυστερούν ακόμα περισσότερα τα παλαιά προγράμματα ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με νέα χρήματα και νέα προγράμματα. Έχετε λοιπόν κάποια πρόταση σε σχέση με το θέμα αυτό. Κατανοώ ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να συμπιεστούν χρονικά, αλλά αυτοί οι οποίοι πληρώνουν τελικά την ύφη είναι οι περιφέρειες και οι δήμοι. Σας ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Κοτσολίνιν έχει το λόγο. Η τελευταία παρατήρηση της Κωνσταντσα είναι πολύ σημαντική. Έχουμε το διτό πρόβλημα στην, σε επίπεδο Ευρώπης. Υπάρχουν χώρες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους 2007-2014 από τη μία. Μπορούμε να σκεφτούμε μία πρωτοβουλία ούτως ώστε να τους επιτρέψουμε να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα χωρίς να χάσουν χρηματοδότηση. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και από την άλλη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καθυστέρηση με την οποία ε, ε, υλοποιούνται οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης, θα οδηγήσουν ε, σε μια καθυστέρηση της ε, έναρξης των προγραμμάτων 2014-2020. Ίσως ξεκινήσουμε το 2015. Μπορεί να έχουμε κάτι, μια καθυστέρηση παραπάνω από κάποιους μήνες. Μπορεί να έχουμε καθυστέρηση δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο. Έχουμε λοιπόν τα, δύο αυτά στοιχεία. Και ακριβώς γι' αυτό είναι σημαντική η παρατήρηση Κωνσταντσα. Γιατί ε, το πρόβλημα είναι πραγματικά περίπλοκο. Και εμείς τις επόμενες εβδομάδε θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα συνειδητοποιήσουμε ότι πολλά προγράμματα ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω στην Ιταλική Προεδρία είναι η εξή. Ίσως δεν έχει φτάσει η στιγμή να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν έχει φτάσει η, η κατάλληλη στιγμή. Από τη μία έχουμε ε, το, το πρόβλημα των ε, δημοσίων επενδύσεων και από την άλλη έχουμε τρομερά αυστηρές προϋποθέσεις για αυτές. Ξεκίνησε μια πρωτοβουλία, νομίζω πέρυσι, από την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων για αυτό το θέμα. Αλλά ποτέ δεν έγινε μια μελέτη, μια εμβάθυνση, ένα σοβαρό προβληματισμό ούτε από το Συμβούλιο ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κόστο που πληρώνουμε εμεί. Γιατί δεν αποσυνδέουμε από την ακαμψία του Συμφώνου Σταθερότητας ε, τους πόρους που η πολιτική συνοχή δίδει στην διάθεση των κρατών μελών. Πόσο, πόση απασχόληση χάνουμε από αυτό. Πόσο ΑΕΠ χάνουμε από αυτό. Εξαιτίας, ας πούμε, όλου αυτού του άκαμπτου πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης. Ας προσπαθήσετε εσείς μαζί με το Κοινοβούλιο να κάνετε ένα προβληματισμό, να ζητήσετε μια μελέτη, ούτω ώστε να αφήσετε στις επόμενες προεδρίες, αλλά και να, στη διάθεση, να έχετε και εσείς στην ε, διάθεσή σας στους επόμενους μήνες, ένα ίχνος, δηλαδή που θα, αποκύπτει, που θα προκύπτει από μια μελέτη. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον προβληματισμό θα καταλάβουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Συχνά εμείς πρέπει να συζητήσουμε για θέματα που δεν τα ξέρουμε καλά για να πάρουμε αποφάσεις με τα λόγου γνώσεως, με την ευαισθησία που, που επιβάλλεται. Ποιο είναι το κόστος της καθυστέρησης της εφαρμογής αυτών των πολιτικών. Πέρα από αυτά τα γενικά νούμερα που μας είπατε, 20% ε, μείωση των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, πόσο κοστίζει σε, με όρους ΑΕΠ, ε, με όρους απασχόλησης, με όρους πολιτικής ε, περιβάλλοντος κτλ. Πόσο κοστίζει αυτό. Έχουμε λίγα στοιχεία για να αποφασίσουμε, για να καταλάβουμε. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν. Αυτό θα μας βοηθούσε για να σκεφτούμε για αυτά τα πράγματα όλοι μας με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Ε, σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Τσίκου. Ευχαριστώ. Συμφωνώ νομίζω με την τελευταία παρέμβαση που άκουσα. Νομίζω κύριε Υφυπουργέ ότι, ότι πρέπει να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση. Θα πρέπει να συνδεθούμε με την πολιτική ανάπτυξης και απασχόλησης, απασχόληση των νέων, αλλά και με τις πολιτικές υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ μπαίνουμε στο θέμα της διαφορετικής μεταχείρισης από περιφέρεια σε περιφέρεια. Η μεγάλη Ευρώπη αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες περιφέρειες. Το 99% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η ραχοκοκαλιά που παράγει, που παράγει ανάπτυξη, που δίνει απασχόληση. Και αυτό το ξεχνάμε. Υπάρχει και μια άλλη διαφορετική μεταχείριση. Ε, η ισότιμη μεταχείριση των φύλων είναι ένα άλλο βασικό θέμα. Και πρέπει να απασχολεί στην πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική του φίλου Που από μελέτε που έχουν γίνει προκύπτει ότι αν υπάρχει ισότητα μπορεί να αυξηθεί το ΑΕΠ. Αν υπήρχε μία εγγύηση ότι υπάρχουν περαιτέρω επενδύσεις, μπορεί να γίνει ένα ποιοτικό άλμα και στην απασχόληση, στην πρόσβαση στην απασχόληση και στην ίση αμοιβή των δύο φίλων. Δεν θέλω να πω περισσότερα σε για άλλα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι η Ιταλική Προεδρία θα πρέπει να κάνει μια παρέμβαση ε, σε αυτό το θέμα. Ούτως ώστε να έχουμε πολιτικές οι οποίες μας επιτρέπουν να ξεπεράσουμε ένα άλλο βασικό δράμα τι σημαίνει για τους νέους, για τις επιχειρήσεις, η διαφορετική πρόσβαση που έχουν νέοι, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι γενικά, στα κονδύλια των ταμείων. Πέρα από την καθυστέρηση των πληρωμών, έτσι. Υπάρχει ήδη πρόβλημα στην πρόσβαση των ταμείων. Είναι ένα τεράστιο δράμα που πρέπει να το ξεπεράσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε και για την επικαιρότητα, όχι μόνο για το μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε τι καλύτερε προποθέσει, ούτω ώστε οι νέοι, οι επιχειρήσει και όλοι όσοι ζουν στο πετσί τους αυτή τη διαφορετική μεταχείριση, να αποκτήσουν την ίδια πρόσβαση. Αυτό είναι για το καλό της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Ευχαριστούμε κύριος Μπόκοβιτς. Ευχαριστώ. Η έκτη έκθεση για τη συνοχή ξεκαθαρίζει πόσο σημαντικά είναι τα κονδύλια της συνοχής για επενδύσεις στις νομιωμένες χώρες μέλη. 20 έως 80% είναι τα ποσοστά των δημόσιων επενδύσεων. Είμαι Σλοβαίνος. Στη Σλοβενία το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων επενδύσεων σε αυτή τη χρονική περίοδο είχε εξαρτηθεί από όρου και συγκεκριμένα από τη χρήση των κονδύλων συνοχής. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το 1 τρίτο του συνόλου των κονδυλίων συνοχής και έχουμε ένα, μια υστέρηση 2007-2011. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της Σλοβενία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Προεδρία πρέπει να βρει μια λύση σε σχέση με τις καθυστερούμενες αυτές πληρωμές, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ολοκληρώσουμε την περίοδο 2007-2011, την περίοδο πληρωμών. Καλό επίσης την Προεδρία να κάνει και ένα βήμα παραπέρα, ώστε όσες χώρες δεν έχουν ακόμη υπογράψει τις συμφωνίες εταιρική σχέσης, να παροτρινθούν να το πράξουν για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Και έτσι στη νέα περίοδο, 2014-2020, να μπορέσουμε να αρχίσουμε να εγκρίνουμε γρήγορα νέα προγράμματα και να αρχίσουμε να αξιοποιούμε τα κονδύλια. Δύο πράγματα λοιπόν. Πρώτον, τι πληρωμές, να λυθεί το πρόβλημα. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη να υπογράψουν τη συμφωνία στο συντομότερο δυνατό. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Έθεριτζ. Ευχαριστώ, θα είμαι σχετικά σύντομος θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ για την τόσο πλήρη παρουσίαση που κάνατε στην αρχή. Ίσως απατώμε, αλλά είπατε ότι θα έπρεπε να αποκλείεται από τα στοιχεία του ελλείμματος η χρηματοδότηση σε επίπεδο συνοχής και πόσο αυτό θα συμβάλλει σε μια πιο υπεύθυνη λογιστική. Κάτι άλλο που είπατε και τον βρήκα ενδιαφέρον. Είπατε για μια προσέγγιση που έχει να κάνει με τα αποτελέσματα. Συμφωνώ μαζί σας. Μα μήπως τελικά αυτό το οποίο προσδοκείται είναι μια κενσιανή διόγκωση των ελλημάτων για να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σας ενδιαφέρει περισσότερο μια συνοχή που θα οδηγήσει σε μια πιο φεδεραλιστική ευρωπαϊκή πολιτική εντότητα. Θεωρείτε ότι τα δύο αυτά στοιχεία συνδέονται και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η απόψή σα για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ, λέγει και η πρόεδρο για τη συντομία σα Και πάλι ο αντιπρόεδρο κύριο Πόλτσακ, έχει το λόγο. σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, έχω ένα πάρα πολύ σύντομο ερώτημα να σας θέσω. σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση των πόρων συνοχής. Η πολιτική συνοχή έχει ένα συνολικό προπολογισμό 150 δισεκατομμύρων ευρώ στο 7 ετές αυτό το πλαίσιο και είναι από τα κύρια στοιχεία υποστήριξη περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξη μικρομεσαίε επιχειρήσει, έχει σαν στόχο να, να μειώσει την ε, ανεργία, υποστηρίζει μια οικονομία χαμηλή χρήση άνθρακο. Το ερώτημα μου το εξή όμω. Εσεί είπατε ότι υπάρχει μια χαμηλή αποτελεσματικότητα για τη χρήση αυτών των πόρων και φυσικά ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε αυτή την αποτελεσματικότητα. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξή. Τι εργαλεία έχει η Ιταλική Προεδρία στη διάθεσή της, τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσει, τι νέα και καινοτόμα εργαλεία θα χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει αυτή την αποτελεσματικότητα των ε, πόρων συνοχής. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Όχι. Κύριε Φίτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Είναι μια έκκληση μετά από τα στοιχεία που ακούσαμε. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να δικαιολογήσουμε τις αρνητικές πρακτικές που υπάρχουν στο εσωτερικό των περιφερειακών πολιτικών. Θα πρέπει να έχουμε και το θάρρος για να παραδεχτούμε κάποιες αποτυχίες, αλλά και για να αξιοποιήσουμε και τις καλές πρακτικές. Το να υπερασπιστούμε απλώς τις πολιτικές αυτές απέναντι στην Κομισιόν θα ήταν λάθος εκ μέρους μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο στοιχεία. Καταρχάς, θέλω να εκφράσω ένα φόβο ότι τα 300 δισεκατομμύρια, τα πολύ γενναιόδωρα, το, το γενναιόδωρο αυτό ποσό για τις μελλοντικέ επενδύσεις, είναι υποτίθεται, όπω λένε οι συνάδελφοι, επιπλέον ποσά. Μακάρι, μακάρι αυτό λέω εγώ, το εύχομαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις πολιτικές συνοχής και τη σημασία του στο, σε επίπεδο προϋπολογισμού. Δεύτερο στοιχείο, δεύτερος προβληματισμός αφορά το σύμφωνο σταθερότητας. Αυτό δεν είναι ερώτημα. Είναι μια έκκληση έντονη, σαφής. Είναι σαφές ότι υπάρχει το πρόβλημα με τις πληρωμές ε, στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2014. Τώρα έχουμε τη νέα περίοδο. Έχουμε παράλληλα το σύμφωνο σταθερότητας και δεν έχουμε, αν δεν δώσουμε απαντήσεις στη σχέση αυτή, τότε θα μας δημιουργηθεί πρόβλημα και σε επίπεδο χρονικό και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και δεν θα δώσουν ανάπτυξη οι επενδύσεις αυτές. Είμαι πεπισμένος ότι εδώ θα έχουμε πολιτικές διαφορές ε, και διαφορές από περιφέρεια σε περιφέρεια. Επαναλαμβάνω κύριε Υπουργέ, δεν είναι ερώτημα αυτό που σας εκφράζω. Είναι μια έκκληση να ληφθούν αυτά τα στοιχεία υπόψη γιατί χρειαζόμαστε ε, σαφείς απαντήσεις σε αυτό το επίπεδο. Thank you, Mr. Fito. now... Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος να που θα ήθελε το λόγο. Όχι, ωραία, ευχαριστώ. Επομένως, ολοκληρώσαμε με τις ερωτήσεις. Στο δεύτερο γύρο, κύριε Ντελρίο, έχετε το λόγο. Μάλιστα. Ακούστηκαν κάποιες ερωτήσεις για την ανάλυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η πρόταση που έγινε από τον κύριο Κοτσολίνο να αξιολογήσουμε το κόστος από επενδύσεις που δεν έγιναν. Ναι, αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε σίγουρα. Δεν έχουμε σκεφτεί αρκετά το κόστος της έλλειψης, της απουσίας επενδύσεων. Τι ανάπτυξη στέρισε, μας στέρισε αυτό στην Ευρώπη. Η δική μας θέση εδώ δεν είναι μια θέση ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε αγνοώντας τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού. Όχι, λειτουργούμε, όπως είπα και στην παρέμβασή μου την αρχική, μέσα σε ένα πλαίσιο που λέει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης να ερμηνευθεί διτά και σε επίπεδο δηλαδή να παίξει το ρόλο του και στη σταθερότητα αλλά και στην ανάπτυξη και να δούμε την επίπτωσή του στο ΕΠ. Εάν γίνει, όπως εμείς ευχόμαστε, επενδύσεις επιπρόσθετες στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, Αυτές τις επενδύσεις θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε και να τις αφαιρέσουμε από, τις, από το σύμφωνο σταθερότητας. Και το ποσοστό συγχρηματοδότησης των διαφόρων κρατών θα πρέπει να θεωρηθεί ε, μια επένδυση απαραίτητη για την ενίσχυση του ΑΕΠ και επομένως είναι μια προσπάθεια πολύ σημαντική. Όπως ξέρετε επίσης γίνονται ήδη διαπραγματεύσεις και υπάρχουν διαδικασίες που επιτρέπουν ε, μια κάποια ευελιξία στη χρησιμοποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την ποσότητα και την ποιότητα των επενδύσεων. Υπάρχει αυτό το στοιχείο. Επίσης προκύπτει σαφώς ότι οι στρατηγικές επενδύσεις, όπως τα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα, οι στρατηγικές επενδύσεις που ενώνουν την Ευρώπη, ούτω ώστε να γίνει μια Ευρώπη ε, ενεργειακά αποδοτική, δημιουργούν, ας πούμε, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο μία πιο σταθερή Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι όμως όλες τι επενδύσεις μπορούμε να τι θεωρήσουμε εξίσου χρήσιμες για την πολιτική ενίσχυση της Ομοσπονδιακής Ευρώπης, όπως είπε κάποιο Ευρωβουλευτή. Η δεν μπορούμε να θεωρήσουμε όλες, ότι όλες αυτές είναι πολιτικές και ε, ενσιανικές για την πρόθεση της απασχόλησης. Πρέπει να αναλύσουμε τις επιπτώσεις αυτών των επενδύσεων. Ε, τι συνέβη με, τα προηγούμενα ε, προγράμματα της περίοδου, προγραμματισμου προγραμματισμού 2007-2014. Έδωσαν διαρκή και μόνιμα αποτελέσματα ή προσωρινά αποτελέσματα. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη εφταετία. θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε τους επόμενους μήνες την διαπραγμάτευση με βάση το αποτέλεσμα του προβληματισμού και να προσαρμόσουμε τα προγράμματα στα αποτελέσματα αυτά. Ωστόσο, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, τους καλύτερους δυνατούς καρπούς. Νομίζω ότι θα μιλήσει γι' αυτό και ο Επίτροπος Χάν που θα με ακολουθήσει. Νομίζω ότι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν την εξάντε ερεσιμότητα. Αυτό είναι σημαντικό για να δουν τι γίνεται με την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Και η δουλειά που έγινε αυτά τα χρόνια για την εξάντε ερεσιμότητα θα βοηθήσει τις επενδύσεις να γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικές. Εδώ θέλω να απαντήσω και στον κύριο Κρέλ. Το θέμα των πληρωμών καταλαβαίνω ότι για σας είναι τα πιο σημαντικά. Ε, επ' αυτού θα πρέπει να εγγύψουμε. Προφανώς. Καταλάβαινα ότι είναι επίγον το θέμα, δεν καταλάβαινα ότι είναι τόσο επίγον. Το καταγράφω και θα, προσπαθώ, θα προσπαθήσω να ασχοληθώ πολύ πιο έντονα με αυτό το θέμα. Όταν όταν φτάσουμε στο τέλος του κύκλου 2007-2013-2014 θα πρέπει να καθυστερήσουν οι πληρωμές. Είναι σαφές. Πάντως νομίζω ότι οι προβλέψεις για τις πληρωμές ε, μπορούμε πληρωμές, στις πληρωμές να βελτιώσουμε τις επιδόσεις αν έχουμε κάνει ε, πολύ καλό προγραμματισμό πριν. Τώρα για τους κανονισμούς. για τα επιχειρησιακά προγράμματα, διορθώνει ο Υφυπουργό. Έχουμε μια καθυστέρηση, γιατί οι κανονισμοί εγκρίθηκαν στο τέλο του 2013, το Δεκέμβριο του 2013. Επομένω τα προγράμματα 2014-2020 θα έχουν μια καθυστέρηση διαφόρων μηνών, αρκετών μηνών, Προφανώ. Σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων πιστεύω ότι ο Επίτροπος Χάν έχει καλύτερες πληροφορίες για να σας δώσει από μένα γιατί παρακολουθεί ο ίδιος προσωπικά αυτά τα θέματα. Κάθε χώρα προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο σε αυτή τη φάση. Και δεν νομίζω ότι το καλύτερο μέτρο, ε, το καλύτερο μέτρο είναι οι αναβολές, οι παρατάσεις, ούτω ώστε να προωθήσουμε τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα. Και το λέω ω εκπρόσωπο μιας χώρας που έχει τον υψηλότερο ε, αριθμό προγραμμάτων κατά απόλυτο τιμή, ε, κατά απόλυτο αριθμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το είπαν και διάφοροι βουλευτέ αυτό, ο κύριος Μπόγκοβιτς λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε αυτή την ε, οδό. Νομίζω ότι συνολικά Μπορούμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις για να τονίσουμε, τονώσουμε τις επενδύσεις. Αυτό που σας ανέφερα στην αρχική μου παρέμβαση, το βασικό σενάριο, η βασική υπόθεση, δεν είναι να έχουμε αποκλεισμού ή να έχουμε γενικές ρήτρε. Ούτε καν ρήτρε αναχώρα. Νομίζω πρέπει να έχουμε μια συνολική στρατηγική, η Κομισιόν δηλαδή, για την ε, επανεκκίνηση της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Και επίσης να δούμε το ποσοστό συγχρηματοδότησης κατά περίπτωση, ακόμα και συνολικά, αφού εγκριθεί, εγκριθούν οι πιο βασικές στρατηγικές επενδύσεις. Και αυτό να αποκλειστεί από τον υπολογισμό του Συμφώνου Σταθερότητας, όπως είπα. Όλες οι εκκλήσεις που έγιναν από τον Τσίτσε, από τον κύριο Κοτσολίνο, από την κυρία Μπρέσο, να δούμε διάφορα σενάρια και από τον κύριο Φίτο. Όλα αυτά τα σενάρια θα πρέπει να τα δούμε αυτούς τους μήνες. Επαναλαμβάνω. Όχι για να αποκλείσουμε επιμέρους χώρες, καθόλου κάτι τέτοιο, αλλά για να έχουμε ένα σφαιρικό πλαίσιο στρατηγικής. Νομίζω ότι με όλα αυτά που σας είπα, απάντησα λίγο πολύ σε όλες τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Μας βοηθήσατε αυτούς τους μήνες που προηγήθηκαν και πιστεύω ότι όλη αυτή η δουλειά ήταν υποφελής για όλους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντελρίο, εξαιρετικά πληροφορική ήταν αυτή η ανταλλαγή απόψεων και στοιχείων. Να υπογραμμίσω ότι όλα τα ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί είναι ουσιαστικά ερωτήματα τα οποία εκπηγάζουν από τον Ευρωπαίο πολίτη. Εκπροσωπούμε τα ερωτήματα που ενδιαφέρουν σε καθημερινό επίπεδο τον πολίτη σε σχέση με την περιφερειακή πολιτική και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Είναι θέματα πληρωμών, αλλά είναι θέματα και εμπιστοσύνης μεταξύ του πολίτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Ελπίζω λοιπόν ότι θα λάβετε υπόψη όλα αυτά τα ερωτήματα και χαιρόμαστε για την παρουσία σας στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Με μεγάλη χαρά θα σας υποδεχτούμε και πάλι εδώ. So have few Ένα σύντομο διάλειμμα για να αποχωρήσει ο κύριος Υπουργός και θα έλθει ο Επίτροπος Χάν. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που μπορώ να καλωσορίσω τον κύριο Ιωάννης Χάν, που είναι ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, ενώπιον της Επιτροπής μας, για την ε, τελευταία, από ό,τι καταλαβαίνω, ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή μας, υπό την τωρινή του ιδιότητα, έτσι δεν είναι κύριε Επίτροπε. Θα δώσω λόγο στον κύριο Επίτροπο για μια σύντομη παρέμβαση. Όχι παραπάνω από 15 λεπτά, ελπίζω. Και μετά θα δώσω το λόγο στους βουλευτές που ενδιαφέρονται να θέσουν ερωτήματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία σας, Επίτροπε Χάν, και σας δίνω το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήλθατε όλοι. Θα ήθελα ιδιαίτερα να χαιρετήσω τον πρώην συναδελφού μου Όλη Ρεν. Πολύ χαίρομαι που είναι στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων και είμαι σίγουρος ότι θα με βοηθήσει στη συνέχεια όταν συζητήσουμε τα θέματα της ε, μακροοικονομικής αιρεσιμότητας και της επιπτώσεις, τους, επιπτώσεις της στην ε, περιφερειακή πολιτική. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, θα ήθελα στην αρχή να μιλήσω γερμανικά, αργότερα αγγλικά. Και πάλι, καλώς ήλθατε όλοι, χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί ξαναβλέπω κάποιους από εσά στα νέα καθήκοντά σας. Και όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, και εγώ υποθέτω θα είναι η τελευταία μου παρουσία ενώπιον σας με την ιδιότητά μου ως Επιτρόπου Περιφερειακών Θεμάτων. Τελευταία ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας. Νομίζω ότι μέσα στα χρόνια που έχουν περάσει και στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή σχέση εργασίας και η ελπίδα μου είναι ότι αυτή η σχέση εργασία μεταξύ της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου θα μπορέσει να συνεχιστεί και στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Πιστεύω ότι μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν που είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Αν θυμηθώ λοιπόν, αν γυρίσω πίσω πέντε χρόνια, θυμάμαι ότι υπήρχαν πολλές αμφιβολίες σε σχέση με την πολιτική περιφερειακών θεμάτων που είχε παρουσιαστεί τότε από την Επιτροπή. Εγώ γνωρίζω ότι η κρίση μας υποχρέωσε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα τα οποία και εγώ υποστήριζα τότε, το θέμα παγκοσχάρη της αντιμετώπισης της ανεργίας και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε αυτή την κοινή προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβάλει αποφασιστικά σε αυτό το εγχείρημα και πολλοί από εσά έχετε δαπανίσει ώρες, βδομάδες, μήνες σε αυτή την προσπάθεια να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή τη συνολική μεταρρύθμιση της περιφερειακής πολιτικής. Πιστεύω όμως ότι έχουμε επιτύχει να συναρμόσουμε καλύτερα την πολιτική αυτή με την πολιτική της Ευρώπης 2020 σε ό,τι αφορά τα θέματα επενδύσεων. Έχουμε λοιπόν ε, ξεκινήσει αυτή την εργασία, αυτό το εγχείρημα μέσα σε μια οικονομική κρίση η οποία είχε πολύ αρνητικά αποτελέσματα για τις περιφέρειες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Από το τέλος του 2012 έχουμε δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του 2012 ότι θα φτάσουμε σε 1,4 ε, εκατομμύρια θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Έχουμε 20.000 ε, περίπου σχέδια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποστήριξή τους, περίπου 80.000 ε, σχέδια για startups, και νέες επιχειρήσεις και έχουμε 60.000 περίπου σχέδια έρευνας και ανάπτυξης τα οποία έχουν δημιουργήσει αντίστοιχα θέσεις στον τομέα της ε, έρευνας και της ανάπτυξης με την υποστήριξη της περιφερειακής πολιτικής. Και όλα αυτά φυσικά έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχουν βοηθήσει πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν μια θέση απασχόλησης. Αυτό φυσικά δεν αλλάζει το γεγονός ότι εξακολουθεί να σοβεί η κρίση στην Ευρώπη και αυτό δεν μας ε, εκπλήσει Ε, στην περίπτωση αυτή ότι έχει αυξηθεί και η ψαλίδα, έχει ανοίξει το χάσμα μεταξύ των ε, πιο προχωρημένων και λιγότερο προχωρημένων περιφερειών στην Ευρώπη. Περίπου 270 περιφέρειες της ε, Ευρώπης είδαν οι επενδύσεις τους να μειώνουν κατά 20% ή περισσότερο και φυσικά και οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν υποστεί περικοπές, οπότε τουλάχιστον το ίμιση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώθηκε να βασίζεται τουλάχιστον κατά 50% στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να φέρει σε πέρας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του. Έχουν φυσικά ε, χρησιμοποιηθεί επωφελώς τα χρήματα αυτά είναι απαραίτητο όμω να υπενθυμίσω την ανάγκη προ όφελο του Ευρωπαίου φορολογούμενου να επενδύονται όλα αυτά τα κονδύλια σε κατευθύνσει, οι οποίε θα είναι παραγωγικέ και θα δημιουργήσουν και ευκαιρίε στο μέλλον. Με την ατζέντα της Ευρώπης 2020 θέλουμε εμεί να συνδέσουμε την στρατηγική αυτή ανάπτυξη με μια εκ των προτέρων εξάντε ερεσιμότητα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει η σωστή εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων και θα μπορούν να συνάδουν με την επίτευξη ποσοτικοποιημένων στόχων. Κατέστη επίσης ε, απαραίτητο να δώσουμε ε, μεγαλύτερη έμφαση στην ε, σύνδεση της περιφερειακής πολιτικής με το ευρωπαϊκό εξάμεινο, ιδίως λόγω της κρίσης η οποία εξακολουθεί να επικρατεί στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε να έχουμε μια καλύτερη ε, μακροοικονομική αξιολόγηση. Εξάλλου έχουμε τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές οι οποίες αναδείχθηκαν σε αυτό το ε, χρονικό διάστημα, όπως αυτή για τις, για τις περιοχές του Δούναβη, για τις περιοχές της Βαλτικής ε, και επίσης με τον τρόπο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα κλίμα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης όπου φαίνεται ο, με τρόπο σαφή ότι υπάρχει μια προσθέμενη αξία η οποία μπορεί να προκύψει από τις ενέργειές μας και μπορούμε να παροτρύνουμε έτσι την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αυτών των περιφερειών και εξάλλου πρέπει να πω ότι και εγώ ίδιος είμαι εντυπωσιασμένος με τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε καταγάγει. Εξάλλου, Έχουμε επιτύχει να φέρουμε την προβληματική των αστικών χώρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι γνωστό ότι 75% ή παραπάνω των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε αστικούς ε, σχηματισμούς, σε πόλεις και μεγάλες κομοπόλεις. Επομένως θέλω και πάλι να το τονίσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως μια συμπληρωματική πολιτική και επομένως δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με μια κατηγορηματική ε, διάκριση μεταξύ πόλεων και περιφερειών και υπέθ, περιοχών της υπαίθρου γιατί είναι αλληλένδετες αυτές. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος σαφής ε, ορισμός που να διαχωρίζει αυτές τις περιπτώσεις αλλά μέσα στην περίοδο προγραμματισμού που έχουμε αντιμετωπίσει είδαμε ότι περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί σε στις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουμε ότι στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 50 ή και 60 δισεκατομμύρια ευρώ θα τεθούν στη διάθεση των πόλεων. Θέλω να σα ευχαριστήσω λοιπόν και όλου αυτού οι οποίοι έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο για να υπάρξει και μία μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύη. κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να χρησιμοποιούμε πιο γρήγορα και να κινητοποιούμε πιο γρήγορα τα κονδύλια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Προφανώς τα κράτη-μέλη έχουν, είχαν, επιβα... επιζητήσει να παραμείνουν αυτά τα χρήματα έξω από, τον, το πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εμείς όμως κάναμε και τις απαραίτητες προσπάθειες για να μπορέσει να μειωθεί και ο χρόνος που χρειάζεται για την εκταμείευση αυτών των κονδυλίων. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου στον ε, αντιπρόεδρό σα και όλους τους συναδέλφους του που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των λύσεων και τώρα μπορώ να γυρίσω στα αγγλικά ίσως. Μπορούμε να πούμε ίσως ότι σε ό,τι αφορά το τι έχουμε πετύχει από κοινού σε σχέση με το όσο είχαμε υποσχεθεί πριν από μια πενταετία περίπου βλέπουμε βέβαια ότι το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης τελικά εντοπίζεται στην υλοποίηση επιτόπου. Υπάρχουν βέβαια ελπιδοφόρα μηνύματα μπορώ να σας πω, αλλά και κάποιες ανησυχητικές ενδείξεις παρόλα αυτά. Παραδείγματο χάρη, κατάσταση ε, υλοποίηση σε σχέση με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. 16 συμφωνίες εταιρικής σχέσης έχουν εκριθεί μέχρι τώρα και κοντεύουμε ε, να κλείσουμε και τις εναπομένουσες. Έχουν υποβληθεί προγράμματα υλοποίησης ε, και σε πολλά έχουμε ήδη διατυπώσει παρατηρήσεις. Επτά όμως μόλις προγράμματα έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα. Οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζουν ενεργά τι ε, διαπραγματεύσει του με τα κράτη-μέλη καθώ και με τι περιφέρειες ώστε να φτάσουμε στο απαραίτητο επίπεδο ποιότητα για μια αποτελεσματική υλοποίηση. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Βέβαια, είμαστε αποφασισμένοι να μην θυσιάσουμε την ποιότητα στο βωμό της ταχύτητας και θέλω να σας το ενθυμίσω και να το τονίσω εκ νέου. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι η ταχύτητα, είναι η ποιότητα. Αν μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο μαζί, ακόμη καλύτερα. Η προτεραιότητά μας όμως είναι η ποιότητα και όχι η ταχύτητα. Μιλάμε για ένα χρονοδιάγραμμα 7, για να μην πω 10 ετών, Άρα νομίζω ότι είναι δικαιολογημένο το ότι θέλουμε να έχουμε έναν υγιή προγραμματισμό για αυτή την περίοδο και στην ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΡΕΚΙΟ αλλά και στις άλλες γενικές διευθύνσεις ε, δεν υπήρξε ε, καλοκαίρι, δεν υπήρξαν διακοπές. Δεν μιλάω για το κλίμα, ότι δεν ήταν καλός ο καιρός. Απλά θέλω να πω ότι όλοι όσοι ε, συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη για τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης δεν έκαναν διακοπές. Ήμασταν λοιπόν διαθέσιμοι, ε, δουλεύαμε όλο το καλοκαίρι και νομίζω ότι το μήνα Αύγουστο σημειώσαμε και σημαντική πρόοδο. Επανέρχομαι τώρα. Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και υπηρεσιακά προγράμματα που έχουν υποβάλει τα κράτη-μέλη. Ήδη Είναι προφανές ότι αποφύγει τους καρπούς της αυτή μεταρρύθμιση. Βλέπουμε μια μετατόπιση σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες χρηματοδότησης. Πολύ ξεκάθαρα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Από τις δικτυακές υποδομές σε τομείς όπως είναι η ενεργειακή απόδοση, ε, μικρές ε, εκπομπές, ε, διοξιδίου του άνθρακα, στήριξη των επιχειρήσεων κτλ. 125 δις ευρώ θα δοθούν για τις βασικές προτεραιότητες του ΕΤΑ και άλλα 100 για το κοινωνικό ταμείο, άρα πάνω από τα 2 τρίτα του προϋπολογισμού συνοχής. Και κάτι ακόμη πιο σημαντικό, πολλά κράτη, πολλές περιφέρειες αποφάσισαν να υπερβούν ε, τις τα κατώτατες ρυθμιστικές απαιτήσεις. Τελικά λοιπόν 37 δις ε, ευρώ περίπου θα ε, στηρίξουν αυτή την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Γιατί προβλεπόντουσαν ως το όριο 23 δισεκατομμύρια από τον κανονισμό. Θα δούμε επίσης να διατίθενται περισσότεροι πόροι σε δάνεια εγγυήσεις και άλλα χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις, επιχορηγήσεις. Ε. Καλό είναι αυτό, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για να έχουμε μεγαλύτερη μόχλευση του κάθε ευρώ που δαπανάται στην πολιτική συνοχή. Υπάρχει κάτι που μας ανησυχεί όμως και θέλω να σας το αναφέρω. Νομίζω είναι η καλύτερη χρονική στιγμή υπό την έννοια ότι είναι καλό το timing. Ο λόγος δεν είναι καλός, τέλος πάντων. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο επίπεδο και στην ποιότητα των δημόσιων επενδύσεων. Αυτό όμως θα πρέπει να συνοδευτεί με μια εξίσου σοβαρή δέσμευση για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών. Στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, στην πολιτική συνοχή, είχαμε καθυστέρηση δηλαδή καθυστέρηση πληρωμών 23,4 δις ευρώ, 23,4 δις, που θα αυξηθεί αυτό ε, το ποσό μέχρι το τέλος του έτους. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τις πιστώσεις πληρωμών για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις δαπάνες για την καινοτομία, για τις ΜΜΕ, για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας, για να μην πω παιδεία, ε, καταπολέμηση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι πιστώσεις πληρωμών που ζητούνται στο σχέδιο διευθυντικού προϋπολογισμού στο τρίτο του 2013 και στο σχέδιο προπολογισμού του 2015 είναι σημαντικές γιατί έτσι θα ε, μειωθεί αυτή η χιονοστιβάδα των ε, ε τιμολογίων και των οργανισμών που δεν έχουν πληρωθεί. Και έτσι θα αποφύγουμε καθυστερήσεις, από πλευρά δικαιούχων και θα στηριχτεί η υλοποίηση των προγραμμάτων. Καλούμε λοιπόν και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τι ευθύνε του. Να αντιμετωπίσουν αυτό το χάσμα, αυτή την αντίφαση μεταξύ των πολιτικών και των θεσμικών δεσμεύσεων από τη μία και τι πληρωμέ από την άλλη. Ολοκληρώνοντα την παρέμβασή μου θα μιλήσω για τι ανοιχτέ ημερίδε, 192 περιφέρειε και πόλει από 31 χώρε και πολλά δίκτυα και ενώσεις σε πάνω από 100 εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις ε, μαζί με 300 τοπικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά θα γίνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη σε δύο εβδομάδες τον Οκτώβριο. Εφής επενδύσεις είναι το βασικό σλόγγαν ε, για όλους. Ο στόχος μας είναι ώστε να το περισσότεροι ευρωβουλευτές να μπορούν να συμμετάσχουν. Πέρυσι δεν κατέστη δυνατό αυτό, ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή τη φορά. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνει η κήρυξη της έναρξης αυτών των ανοιχτών ημερών και για πρώτη φορά αυτό θα συνοδευτεί και με κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ρέγγι και Κότερ και έτσι θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες συζήτησης με ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία διοικητικών υποδομών, διαφορετικά ταμεία, ταμείο συνοχής και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε και τους δύο Προέδρους Επιτροπής Περιφερειών, την κυρία Μπρέσο και τον κύριο Βαλκάρθελ. Θέλω να τους ευχαριστήσω προσωπικά και εμένα και όλους τους ε, συναδέλφους μας συνόδευσαν στην προηγούμενη πενταετία και έχουν σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία της πολιτικής συνοχής. Θέλω λοιπόν να σας ε, ενθαρρύνω, να σας πατρύνω να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτές τις ανοιχτές ε, ημέρες και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νέα Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει και την πρότασή της για το πολιτές πλαίσιο. Ελπίζουμε η Επιτροπή σας να συμμετάσχει ήδη από τώρα, έστω στο τέλος αυτής της εντολής, για τη συζήτηση και για την προετοιμασία. Ελπίζω να βοηθήσετε να προετοιμάσετε και το διάδοχό μου για το έργο που έχει να λαλάβει τις επόμενες χρονιές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λάβουμε πολλές πληροφορίες. Ακούσαμε μία περίληψη των επιτυχιών σας, αλλά και των προβλημάτων που εξακολουθούν να σοβούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις πληροφορίες. Έχουμε 45 λεπτά για συζήτηση, για ανταλλαγή απόψεων. Και να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις των συντονιστών. Ο κ. Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ η παρουσία του κυρίου Χάν ε, δεν συνιστά ακρόαση, αλίμονο. Το να κάνουμε ερωτήσεις δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Ε, σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε τον κύριο Χάν, κάναμε ερωτήσεις. Είχαμε θαυμάσιο διάλογο, επικοδομητικό. Αν συνειδητοποιήσετε από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε, όλη αυτή η ολοκληρωμένη πολιτική Συνοχή και περιφερειακή πολιτική δεν ήταν κάτι το δεδομένο στην αρχή. Υπήρχε τάση, μάλιστα, να τα βλέπουμε τα πράγματα ε, κατακαιρματισμένα. Χρηματοδότηση για την ενέργεια από τη μία, από την άλλη χρηματοδότηση άλλων πολιτικών της ε, Ευρώπης 2020. Κατακαιρματισμένα όμως. Και τι προέκυψε μετά από όλη την προσπάθεια, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική, όπου οι μεγαλύτερες επενδύσεις προέρχονται από τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθωτικών Ταμείων και, του... και Επενδυτικών Ταμείων. Είναι σαφές λοιπόν ότι υπάρχει μία πρόοδος εδώ, όπως προκύπτει και από την έκτη έκθεση. Αυτή είναι η κληρονομιά σας, αυτά κάνατε. Uh, Επίσης συνδυάσατε πολύ καλά τα, αυτά τα κονδύλια με τα, ταμεία έρευνα, κονδύλια από το Ταμείο Έρευνας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στα ΜΕΝ και στα ΔΕ ε, συνεργάζονται τώρα καλύτερα, ούτως ώστε να έχουν μια πιο έξυπνη, πιο πράσινη Ευρώπη, με προσανατολισμό στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σας ευχαριστώ για αυτό. Κάτι που δεν κατάλαβα από αυτά που είπατε. Ξέρω ότι είσαστε από τις Άλπεις, από μια περιοχή της, της Άλπης. Μιλήσατε για μια χιονοστιβάδα ε, ή για μια επίπτωση έτσι, τύπου snowboard. Γιατί οι επιπτώσεις της ε, ανεπαρκούς ε, πληρωμής μπορεί να είναι είτε χιονοστιβάδα είτε επίπτωση snowboard. Ε, δεν είμαι καλό αλλά μπορεί να είναι το ένα ή το άλλο. Η συνάδελφό σα, κυρία Γκέγκελ, ήρθε στην Ολομέλεια και είπε τι προάλλε ότι αν δεν ε, βελτιωθεί η κατάσταση των πληρωμών, το 2020 θα φτάσουμε σε μια έλλειψη πληρωμών ύψου 40%. Ας το δούμε έτσι, όπως είναι. Ίσως μπορούμε να αποφύγουμε λοιπόν τη χιονοστιβάδα σε αυτό το επίπεδο. Τώρα πιο σοβαρά. Το ΕΛΚ σας ευχαριστεί πολύ για τη δέσμευσή σας και για τη νομοθετική δουλειά που κάναμε, τη δουλειά που κάναμε σε επίπεδο κανονισμών και όλη την ε, συμβολή σας σε κάθε χρονική στιγμή. Δεν είμαστε πάντα αντίπαλοι εμείς η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Πολύ συχνά ήμασταν, ε, δώσαμε τη μάχη μαζί. Συχνά στρέφομαι προς τους εκπροσώπους του, Συμβουλίου και αυτοί είναι στη, μεριά, στη γωνιά τους. Ε, αυτή είναι η αντιπαλή μας στους διάφορους τριμερείς διαλόγους. Ε, είχαμε περίπου 150-200 τριμερείς διαλόγους. Ε, για ένα κανονισμό από αυτούς είχαμε μόνο 80 τριμερείς διαλόγους. Ε, αυτά κάναμε το παλιό κοινοβούλιο. Ελπίζω το νέο κοινοβούλιο να συνεργαστεί και να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα ερωτήματα που μας θέτουν οι διαδοχικές κρίσεις. Ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια σταθερή βάση για ανάπτυξη, καλές σχέσεις ανάμεσα στις ε, περιφέρειες, τα κράτη και όλους όσους δραστηριοποιούνται στα διάφορα επίπεδα. Ευχαριστούμε κύριε Νίστλερ. Η κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, Χάν, νομίζω ότι εξ ονόματος όλη τη σοσιαλιστικής ομάδα μπορώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε εσά για τον χρόνο που ήσασταν ο επίτροπο για τα περιφερειακά θέματα, για όλο τον χρόνο που περάσαμε μαζί, για την κοινή εργασία που κάναμε μαζί, για την διαθεσιμότητά σας ακόμα και όταν η Κομισιόν δεν είχε την ίδια άποψη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρόλα αυτά να συζητήσετε μαζί μας, να παρουσιάσετε στοιχεία και επιχειρήματα υπέρ της δικής μας θέσης. Αυτό ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία στις διαπραγματεύσεις που είχαμε. Το γεγονός ότι εσείς πάντα λαμβάνετε την άποψη των άλλων. και ήταν πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πόση ικανότητα πολλές φορές μπορεί να συγκεντρώσει το Συμβούλιο και η Κομισιόν σε επίπεδο τεκμηρίωσης και εργασίας και εμείς ως Κοινοβούλιο πολλές φορές με λιγότερα υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό στην, στη διάθεσή μας αναγκαστήκαμε και εμείς να επομιστούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βάρος σε επίπεδο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και τεκμηρίωσης και εκεί μας βοήθησε η Κομισιόν και μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να επιτύχουμε ένα μεγάλο μέρος από τους στόχους μας, όχι πάντα, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική η υποστήριξη της Κομισιόν και Μον με Νομίζω επίσης ότι έχετε αφήσει κάποιες ανοιχτές ε, πόρτες σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της πολιτικής έρευνας και της ε, εκμετάλλευσης έρευνας για να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή επίσης για ζητήματα των προβλημάτων που έχουν να κάνουν οι πόλεις και πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αηφόρο ανάπτυξη και εξέλιξη των πόλεων ή επίσης σε ό,τι αφορά το θέμα της δημογραφικής αλλαγής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό εδώ και πάρα πολύ καιρό αλλά είναι ελάχιστες οι απαντήσεις οι οποίες έχουν δοθεί για το θέμα αυτό και στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν υπάρξει κάποιες περισσότερες προσπάθειες ώστε να δημιουργηθεί μια πολιτική συνοχής η οποία να συνδέει πραγματικά τις περιφέρειες της Ευρώπης και μπορεί να αντιμετωπίσει τα απτά προβλήματα των ανθρώπων στην Ευρώπη. Και έρχομαι τώρα σε κάποια ερωτήματα. Σε πολλές συζητήσεις, τριγωνικούς διαλόγους, διαπραγματεύσεις, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα πακέτο για τη νέα πολιτική περιφερειακών θεμάτων και εμείς ως Κοινοβούλιο ίσως δεν έχουμε περατώσει εγκαίρο την επεξεργασία μας. Είναι σαφές όμως ότι δεν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα σε σχέση με την εφαρμογή μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Ανησυχώ όμως παρόλα αυτά λιγάκι όταν βλέπω ότι υπάρχουν 16 συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης μονάχα και 7 περαιτέρω προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την ε, Κομισιόν. Φυσικά δεν φταίει η Κομισιόν, φταίνουν τα κράτη-μέλη που δεν έχουν κάνει την απαραίτητη προπαρασκευαστική εργασία. Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να επιταχύνουμε κάπως και να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία. Γιατί μας ενδιαφέρει τα μάλα, το ταχύτερο δυνατό να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα λειτουργικά προγράμματα στις περιφέρειες της Ευρώπης και με τον τρόπο αυτό να μπορέσουν οι πολίτες και οι πολίτησες της Ευρώπης να διαπιστώσουν ότι πράγματι το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει και μας νοιάζει ιδιαίτερα να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των περιφερειών και ότι έχουμε δημιουργήσει ένα οπλοστάσιο μέτρων τα οποία μπορεί να βοηθήσει τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να έχω κάποιες ενδείξεις από τη δική σας πλευρά κατά τόσο, κατά τόσο κατά πόσο ισχύει αυτό. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο σημείο, λέτε ότι είναι πιο σημαντική η ποιότητα από την ταχύτητα, αλλά υπάρχει κάποια δυνατότητα να ενταπιστούν κάποια προγράμματα ποιότητας τα οποία να μπορούν να προωθηθούν και ακόμα και δεν έχει εγκριθεί πλήρως το λειτουργικό πρόγραμμα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των περιφερειών και να πούμε ότι ξεκινάμε τις διαδικασίες και όταν πράγματι εγκριθεί θα μπορέσει να τύχει της πλήρους χρηματοδότησης από τα διαφορετικά ταμεία ώστε να μην δημιουργηθούν χάσματα και κενά και να μην χρειαστεί να διακοπούν αξιόλογα προγράμματα τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να επανεκκινήσουν. Γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω την ευαρέσκειά μου αν μπορούμε μέσα στα πλαίσια αυτής της τελευταίας επίσημης επαφής με εσά να έχουμε το μήνυμα ότι πράγματι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες να δοθούν κάποιες μεταβατικές λύσεις υπέρ των περιφερειών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κρέλ. Κύριε Νίκολσον, θέλετε να λάβετε το λόγο. Όχι. Κύριο Γιακουβτσίτς. Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι μέχρι πρόσφατα καθόμουν από την άλλη μεριά του τραπεζιού και χρησιμοποιούσα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ήμουν περιφερειάρχη σε μια περιφέρεια της Κροατίας μέχρι πρότινος. Πρέπει να σας πω λοιπόν ποια ε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μικρά και μεγάλα προγράμματα. Και προώθησα καμία εκατοστή προγράμματα, πρέπει να σας πω, που χρηματοδοτήθηκαν και με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με συγχρηματοδότηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν ως πρώην Περιφερειάρχης για αυτή τη συνεργασία και ελπίζω η συνεργασία να συνεχιστεί και στο μέλλον. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για ένα, ε, για ένα πρόβλημα που υπάρχει. Δύο μάλιστα, όχι ένα μόνο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε καταρχάς κάποιες διαδικασίες. Ειδικά για κάποια έργα τα οποία ξεκινάνε τρέχουν και μετά ξαναρχίζουν πάλι. Μιλάμε για, για έργα τα οποία μοιάζουν με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βρούμε κάποιους, κάποιες εύκολες λύσεις για να βοηθήσουμε στη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Ε, μιλάμε καμιά φορά για καλά προγράμματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί στο παρελθόν, ήταν καλά, απέδειξαν την αξία τους και χρηματοδοτήθηκαν στο παρελθόν. Να σας μιλήσω και ένα, πρόγραμμα που έχουμε, ένα πρόβλημα που έχουμε ε, στην υλοποίηση προγραμμάτων μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης από πλευράς της ε, σλοβενικής εθνικής εκπροσώπησης. Μερικές φορές ε, μας μπλοκάρουν οι Σλοβαίνοι μήνες ή και ένα χρόνο. Δεν, ε, δεν είναι θέμα χρημάτων, έχουμε τα λεφτά. Μερικές φορές δεν υπάρχει, δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις. Χρειάζεται και μια οργάνωση, έτσι, σε επίπεδο επιχειρήσεων στο μη κρατικό τομέα. Έτσι. Μπορείτε να, δείτε, να πάτε να δείτε τι γίνεται με τους γειτονέ μας. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους, ε, την πλευρά αυτή να λάβουν ε, αποφάσεις. Ε, γιατί και οι περιφέρειες και οι επιχειρήσεις έχουν επενδύσει σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτά τα προγράμματα, όλα αυτά, οι δικές μας επιχειρήσεις, εντάξει, αλλά εξαιτίας της καθυστέρησης της Λουμπλιάνα κολλάμε κι εμείς, είμαστε στον τοίχο. Τώρα, για τη μελλοντική σας δουλειά θέλω να πω κάτι. Ξέρετε ότι είχαμε όλες αυτές τις ε, φοβερές πλημμύρες στην Κροατία και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Καλό θα ήταν να μπορέσετε κι εσείς να δείτε τι γίνεται εκεί πέρα, να βοηθήσετε, να επισκεφθείτε τις περιοχές που πλημμύρισαν και να δείτε τι συνέβη. Σας ευχαριστώ. Θα το λόγο στον Αντιπρόεδρο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω και εγώ να τονίσω την καλή σχέση που υπήρχε μεταξύ της Επιτροπής μας, της διαπραγματευτικής μας ομάδας, κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Επιτρόπου Χαν όλος ιδιαιτέρως. Μας ακούγατε πάντα, ακούγατε τις απόψεις και τα αιτήματα των Ευρωβουλευτών και σας ευχαριστώ για αυτό. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την ιδιαίτερη προσοχή που δείξατε στις ε, υπερπόντιες και υπερπεριφερειακές περιοχές. Ήρθατε, τις επισκεφτήκατε και στην ε, Ρεουνιόν και στη Μαγιότ και ελπίζω αυτή η νέα πνοή που δώσατε να μην σταματήσει εδώ με την αποχώρησή σας. Είχαμε πάνω από 100 συνεδριάσεις στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου για να προσαρμόσουμε τελικά τα ταμεία συνοχής στις νέες προκλήσεις. Σε ένα κόσμο που αλλάζει όλο ένα. Τα διαφθορτικά ταμεία, χωρίς το Ταμείο Αλληλεγγύης πια. Επιτρέψαμε να γίνουν ταμεία όμως για τις επενδύσεις προσαρμοσμένα στις νέες προκλήσεις, που είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα, η κλιματική αλλαγή, προβλήματα στις αστικές περιοχές κτλ. λοιπά. Και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Παραδείγματος χάρη να προβληματιστούμε για τις στρατηγικές, τις περιφερειακές προσαρμογής απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Είπατε ότι πάνω από 70% του πληθυσμού ζει στις πόλεις. Αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς να εμπλέξουμε πολύ πιο έντονα και τις πόλεις και τις περιφέρειες. Νομίζω όμως ότι στην ουσία σώσαμε τα πιο βασικά πράγματα που είναι η βασική αρχή της ε, περιφερειακής πολιτικής μέχρι το 2020. Θα πρέπει τώρα να σκεφτούμε τι γίνεται μετά το 2020. με δεδομένα περίπλοκα, το ξέρουμε, με πολιτικά δεδομένα που είναι εξελίξη και ρευστά, με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και μια και είσαστε συνυπεύθυνο αυτών των κανονισμών σε αυτή τη διαπραγμάτευση, έχουμε τώρα πια την συνυπευθυνότητα να υλοποιήσουμε το κανονισμό αυτό μέχρι την ε, παραμονή των νέων διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε η νέα πολιτική να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην σας πω περισσότερα, αλλά να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την σχέση αυτή που δημιουργήσατε, την εταιρική σχέση αυτή που δημιουργήσατε. Κυρία Βαν. Σας ευχαριστώ. Είμαι νεότευκτη σε αυτή την Επιτροπή και σε αυτό το Κοινοβούλιο, κύριε Επίτροπε Χάν. Σας ξέρω από το παρελθόν βέβαια στην δημοτική πολιτική της ε, Βιέννης. Βρεθήκαμε βέβαια σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τα θέματα αυτά, αλλά παρόλα αυτά εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τον ρόλο που παίξατε ως Επίτροπος για τα περιφερειακά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι έχετε βοηθήσει ιδιαίτερα στην αξιοπιστία αυτής της πολιτικής και ιδίως για την πολιτική που έχει να κάνει με τον αστικό χώρο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι και αυτό έχει βοηθήσει και την πόλη μας στη Βιέννη να προχωρήσει λίγο περισσότερο. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν παρά να αντιμετωπιστούν θετικά γιατί έχουν βοηθήσει και την οικονομική και ε, κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας έχει βοηθήσει να ξεπεράσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κρίση όπως λέει και η έκτη έκθεση για την περιφερειακή πολιτική. Παραμένει βέβαια το θέμα της ε, παροχής ε, θεμελιωδών δημοσίων υπηρεσιών που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στο μέλλον και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση, ε, να συνεχιστεί η ενέργεια αυτή από τη βάση αυτών που έχετε επιτύχει εσείς τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχετε μιλήσει για 50 δισεκατομμύρια επενδύσεων για τις πόλεις. Φυσικά αυτό είναι σταγόν εν το ωκεανό και πράγματι η πολιτική συνοχής πρέπει να γίνει αντιληπτή ως πολιτική επενδύσεων. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα αυτές οι επενδύσεις. Ξέρουμε ότι πάρα πολλές πόλεις δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τις επενδύσεις αυτές λόγω των περιορισμών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ξέρετε λοιπόν ότι υπάρχει αυτός ο περιοριστικός χαρακτήρας του Συμφώνου Σταθερότητας. Και επομένω δεν μπορούν οι πόλει να κάνουν τι απαραίτητε επενδύσει ώστε να προωθήσουν τους στόχους της Ευρώπης 2020 που αναφέρατε και εσεί. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξή. Στην παραταξιακή ομάδα για τι δημόσιε υπηρεσίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε μια πρόταση η οποία διατυπώθηκε να υπάρχουν επενδύσεις για τις ε, δημόσιες επενδύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ιδίως να αφαιρεθούν από τον υπολογισμό του ελλείμματος <clears throat> και συζητήσαμε ήδη με τον εκπρόσωπο της Ιταλικής Προεδρίας ώστε να αφαιρεθεί, για τη δυνατότητα να αφαιρεθεί αυτή η συγχρηματοδότηση από τα κριτήρια για το δημόσιο έλλειμμα. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε ποια είναι η θέση σας για τις μακροπρόθεσμες αυτές επενδύσεις, ιδίως στους Δήμους και τις κοινότητες που έχουν χαρακτήρα μακροχρόνιων επενδύσεων υποδομών η κυρία Μαρίτα. Νταμάτο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο. Ποια, με βάση την παρελθούσα εμπειρία σας, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις, αλλά και σε εμά και στο νέο Επίτροπο, για τα συστήματα ελέγχου των ε, εξόδων, χωρίς να φτάσουμε σε επίπεδο καταγγελιών, όπως κάνει η Όλαφ, που φέρνουν άλλα αποτελέσματα. Εμείς άλλο ζητάμε. Είδαμε ότι πολλά κράτη ε, είναι καθυστερημένα στην παρουσίαση των συμφωνιών εταιρικής, σκέψης, ε, εταιρικής σχέσης. Έχετε κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν να επιταχύνουν τη δουλειά τους στα κράτη-μέλη αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του Ευρώπη 2020. Το λέω για να βοηθήσουμε αυτά τα κράτη, για να ετοιμαστούν. Γιατί είναι σημαντικό και το χρονοδιάγραμμα ε, για τον τρόπο μοιράσματο των ε, κονδυλίων των ταμείων. Επίσης, μια στρατηγική ε, μετατροπής της ε, βιομηχανίας. Να ξεφύγουμε. Επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα, ε, έχουμε εγκαταλείψει τις πολύ βαριές παραδοσιακές βιομηχανικές δομές και κινούμαστε προς ε, μια κατεύθυνση πιο ευνοϊκή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Τελειώσαμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας λόγια. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να συνενώσουμε τα θετικά στοιχεία που είχαμε ο καθένας από μας. Και είμαι πεπισμένος ότι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου ε, θα μπορέσουμε μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας με την ε, σε τρέχουσες επιτροπής θα μπορέσουμε να ε, λύσουμε όλα τα θέματα με, τις, με τα κράτη-μέλη εκτός της Κροατίας που θα καθυστερήσει ενδεχομένως λίγο περισσότερο λόγω των προβλημάτων που αναφέρθηκαν και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την έγκριση των λειτουργικών προγραμμάτων που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί. Προχωρούν τα πράγματα λοιπόν διαδοχικά. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι τα προγράμματα αυτά εταιρικού χαρακούν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Σπάνε τα, τη λογική των στεγανών που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν. Επιτρέπει να δούμε περισσότερο ποιες ευκαιρίες έχουμε για να προωθήσουμε τα πράγματα αυτά χωρίς να είμαστε στα παραδοσιακά πλαίσια και αυτό σημαίνει και για τα κάτι μέλη ότι απαιτείται μια περαιτέρω συνεργασία και συντονισμός μεταξύ Υπουργείων και μεταξύ Περιφερειών. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει βοηθήσει και σε επίπεδο ποιότητος, αλλά μπορούμε να είμαστε εξίσου ικανοποιημένοι και από την ταχύτητα με την οποία έχουν επιτευχθεί αυτά σε χρονικό επίπεδο. Βέβαια, στα κράτη-μέλη υπάρχει κάποια, κάποια τάση να μην θεωρούν ιδιαίτερα θετική αυτή την έννοια της ευκαμψίας. Και αυτό μας υποχρέωσε στο να έχουμε μακροσκελείς συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για τα ζητήματα αυτά. Κάτι ακόμα για το οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας και σας ε, παρακαλώ να το εξετάσετε αυτό και ενδεχομένως μπορούμε να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες σε διμερές επίπεδο για συγκεκριμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πολιτική για τα διάφορα σχέδια τα οποία πρέπει να εφαρμόσουμε και αυτό δεν έχει περάσει ως μήνυμα ακόμα στα κράτη-μέλη. Σε πάρα πολλούς τομείς λοιπόν έχουμε ακόμα την ανάγκη να υπάρξει μια στρατηγική από τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να γίνει κατανοητό με ποιους στόχους θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους πόρους και να συμφωνήσουμε με τα κράτη-μέλη στρατηγικές ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα στα εγχειρήματα αυτά. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο νέος επίτροπος ή η νέα επίτροπος θα μπορέσει και αυτή να συμβάλλει στην συζήτηση αυτή και φυσικά θα πρέπει να πριτανεύουν και εκεί στη συζήτηση αυτή οι αρχές της ποιότητας και της ε, αν δείτε τώρα τα θέματα των πληρωμών, το ρεύμα πληρωμών που πηγαίνει στα κράτη-μέλη, εφέτος και του χρόνου θα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό πληρωμών που θα αφορά ακόμα το χρονικό διάστημα 2007-2013 και που σε ορισμένε περιπτώσεις θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να περατωθούν πλήρως μέχρι το 2015. Από το επόμενο χρόνο, εγώ θεωρώ ότι θα μπορέσει να γίνει δυνατό να καταβάλουμε τις πρώτες πληρωμές για προγράμματα της περίοδου προγραμματισμού 2014-2020. Και θα πρέπει φυσικά να δούμε ότι θα υπάρξει μια επικάλυψη αυτών των δύο χρονικών περιόδων σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. και φυσικά μπορούν να ξεκινήσουν αυτά τα ερωτήματα που μου απευθύνθηκαν. Μπορούν οι περιφέρειες και οι χώρες να ξεκινήσουν με νέα προγράμματα, ακόμα και εκεί που δεν έχουν συναυτεί οι απαραίτητες ε, συμφωνίες. Πιστεύω λοιπόν ότι κατά 90%, κατά 95% θα μπορέσουν τα προγράμματα αυτά τα οποία υπάρχουν μορφή απλώς προσχεδίου θα μπορέσουν πιστεύω να ε, γίνουν δεκτά και έτσι έχουμε ήδη μια πολύ καλή σχέση με τους ε, εμπειρογνώμονες των περιφερειών και μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία προγραμματισμού θα μπορέσει να συνεχίσει με ομαλό τρόπο και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα υπάρξει κανένα πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί και εν γέννη γνωρίζετε πολύ καλά όπως και εγώ ο ίδιος πού βρίσκονται τα προβλήματα σε κάθε χώρα ή σε κάθε περιφέρεια θα πρέπει κάθε φορά να εξασφαλίζουμε το ότι θα περατωθεί με τακτικό τρόπο η χρονική η περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 και να μην αφήσουμε κονδύλια τα οποία θα παραμείνουν εκρεμή. Ε, δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος αυτός στην τρέχουσα αυτή περίοδο η οποία περαιτώνεται, διότι η ποιότητα της διοίκησης της περιφέρειας αυτές έχει βελτιωθεί και έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν μια πραγματική σταθερότητα σε ό,τι αφορμογεί τα κονδύλια αυτά. Και επανέρχομαι τώρα στην συνοχή Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να διευκολύνουμε και να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Μπορούμε να πούμε ότι ελοχεύει ακόμα ο πειρασμός στα κράτη-μέλη να έχουν περαιτέρω στρώσεις μέσα σε εισαγωγικά απαιτήσεων, αυτό το οποίο ονομάζουμε στα αγγλικά gold plating. Έχουμε προσπαθήσει και εμείς να εφαρμόσουμε την αρχή του ενιαίου λογιστικού ελέγχου, το οποίο σημαίνει ότι εφόσον αυτό είναι εφικτό, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη αξιοπιστία ότι η ποιότητα της, ε, του λογιστικού ελέγχου, αν η ποιότητα του λογιστικού ελέγχου είναι δεδομένη, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε και εμείς τους ε, ελέγχους που κάνουμε σε επίπεδο τελικού δικαιούχου, ώστε να βελτιώσουμε τη διαδικασία και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ε, σχέδια, έχουμε την διαρθρωμένη αυτή διαδικασία που θα επιτρέψει στους ετούντες να χρησιμοποιήσουν τις δομές αυτές που επιτρέπουν μια σωστή προετοιμασία των μιζώνων σχεδίων και στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές θα είναι δυνατό η Κομισιόν να βασίζεται σε αυτές τις ε, ε, κρίσεις που έχουν γίνει για τις ε, διαδικασίες και θα χρειαστεί να έχουμε μια πρόσθετη ε, διαδικασία αξιολόγηση, όλα αυτά θα μπορέσουν να επιταχύνουν για ορισμένα σχέδια τη διαδικασία αξιολόγηση. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία των αξιολογήσεων σε σχέση με τις ε, αιτήσει που έχουμε λάβει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης από την Κροατία, αλλά και από τη Σερβία, την Βοσνία-Σεγοβίνη που δεν εμπίπτουν μέσα στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης. Υπήρξαν όμως και άλλες ευκαιρίες, υπήρξε μια συνδιάσκευση χορηγών που θα μπορέσει να δώσει 800 εκατομμύρια ευρώ στη Βοσνία Ζεχοβίνη για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις ε, φυσικές καταστροφές που έλαβαν χώρα και να επισκευάσει και να ε, βελτιώσει την, ε, τις υποδομές της που κατεστράφησαν. Έρχομαι τώρα στο θέμα των πόλεων. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν. Όπως ελέγχθη, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020, θα πρέπει να στοιχηματίσουμε στις πόλεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ για το ενδιαφέρον αυτό πείραμα που έγινε στην Ιταλία με τη δημιουργία μητροπολιτικών δομών. Αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν όλα αυτά να εφαρμοστούν στην πράξη επωφελώς. Και για τα μέτρα επενδύσεων παραμένει να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν έχει κάθε χώρα το ίδιο συνταγματικό πλαίσιο. Τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτικά στην οργάνωσή τους εντάξει έχουμε και την Ιταλία, την ε, ε, Αυστρία και την Ισπανία που ίσως αποτελούν εξαιρέσεις, αλλά υπάρχουν κανόνες παραγωγός χάρη σε βατικές χώρες ή στην ε, Γαλλία, βάσει των οποίων οι Δήμοι δεν έχουν το δικαίωμα να <clears throat> αναλαμβάνουν να, να είναι δανειολήπτες, να συνάπτουν χρέη. Οπότε αυτό επηρεάζει το θέμα της <clears throat> μακροοικονομικής ερεσιμότητος. Και είναι κατά κάποιο τρόπο οι δήμοι αυτοί και οι κοινότητε θύματα της συνολικά αρνητικής μακροοικονομικής απόδοσης των χωρών τους. Και στην Ιταλία νομίζω ότι υπήρξε αυτή η δυνατότητα να εφαρμοστεί η ρήτρα αυτή επενδύσεων, η οποία επιτρέπει να υπάρξουν επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από ε, κονδύλια συνοχής να μην υπάρχει αυτή η πρόταση να μην περιλαμβάνονται στα κριτήρια του Μάστριχτ. Είναι απαραίτητο εδώ τα κράτη-μέλη να βρούνε μια κοινή θέση γιατί υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες για το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω φυσικά ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα Κατανοώ φυσικά και τις δυσκολίες οι οποίες θα συνδεόντουσαν με μια τέτοια προσέγγιση. Και θα υπήρχαν προβλήματα εάν υπήρχε μια ιδιαίτερα διασταλτική ερμηνεία του τι σημαίνουν ε, επενδύσεις για ορισμένα σχέδια. Όπως είπα λοιπόν, μπορώ να το πω τηλεγραφικά ότι η πρόθεση είναι κάτι το οποίο μπορώ να το κατανοήσω απόλυτα, αλλά ο, διάβολος ως είναι γνωστό κρύβεται μεταξύ των λεπτομεριών και θα πρέπει ενδεχομένως να εξασφαλίσουμε ότι δεν ξεπερνάει κανείς με τις δημόσιες επενδύσεις ένα πολύ μεγάλο επίπεδο κονδυλίων. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί την ε, έγκριση των κρατών μελών και θα έλεγα ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο σε εγχειρήματα τα οποία υπάρχουν ήδη και αυτά είχαν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν με μια πρωτοβουλία του συναδέλφου μου, του τότε συναδέλφου μου Όλη Ρεν, μια πρωτοβουλία που έδινε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την δυνατότητα η οι επιδοτήσεις που δίδονται από διαφορετικά ταμεία προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρηματοδοτούνται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε να μην χρειάζεται καθόλου εθνική συγχρηματοδότηση. Όταν βλέπω λοιπόν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ευρώπης προβλήματα πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση, το μόνο το οποίο μπορώ να κάνω είναι να σας ε, προσκαλέσω να ξανασκεφτείτε αυτή τη δυνατότητα που είχε δημιουργηθεί να υπάρχουν πρωτοβουλίες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να μπορούν να χρηματοδοτούνται 100% από ενωσιακά κονδύλια χωρίς να έχουν απέτηση εθνικής συγχρηματοδότησης. Και προς τη συνάδελφο από την Ιταλία, μια τελική παρατήρηση, χρειαζόμαστε και τη βιομηχανία και χρειαζόμαστε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι χρήσιμο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να έχει τεχνολογίες εχμής και είναι χρήσιμο να σκεφτούμε περισσότερο για αυτές τις τεχνολογίες εχμής ή τεχνολογίες κλίδια πώς θα μπορούσαμε να τις ε, ενισχύσουμε όχι μονάχα σε επίπεδο χρηματοδότηση, αλλά δημιουργώντα και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα να τα αξιοποιήσουμε. Who... Έχουμε και τον κατάλογο των συναδέλφων που θέλουν να θέσουν ερωτήσει στον Επίτροπο. Σας ζητώ να είσαστε πολύ λακωνικοί για να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε όλου. Κύριο Ζέλα. Ξέρω ότι έχετε λίγο χρόνο. Έχω πολλά να πω βέβαια, αλλά θα σταθώ μοναχά σε τρία ή τέσσερα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Επίτροπο Χάν για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στο παρελθόν. Πολλοί θεωρούσαν ότι η Κομισιόν είναι πιο κοντά στο Συμβούλιο, αλλά εσείς χρησιμοποιήσατε και την συνδίκη της Λισαβόνας για να δείξετε το σεβασμό που έχετε προς το Κοινοβούλιο και το γεγονός ότι είστε πιο κοντά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξαν οι συνέπειες αυτές που αναφέρατε για την αστική πολιτική, την πολιτική των αστικών χώρων που συμπεριλαμβάνεται και αυτή στο χώρο της περιφερειακής πολιτικής. Τα κατανοούμε αυτά. Το ερώτημα είναι πόσο σοβαρά θα ληφθεί αυτό υπόψη στην εφαρμογή. Εμείς αγωνιστήκαμε για να υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας για τα κράτη-μέλη, αλλά και εσείς από τη δική σας πλευρά θα πρέπει να εξασφαλίσετε να αναγνωρίσετε την πολυεπίπεδη πολιτική και γνωρίζω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε όλα τα κράτη-μέλη και ιδίως στα μικρότερα στους μικρότερους, ε, μικρότερες πόλεις παραμένουν προβλήματα με την χρηματοδότηση Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους να διαχωρίσουν τα επίπεδα διακυβέρνησης. Και υπάρχει επιπλέον το θέμα του προπολογισμού. Ο jean Κλωτ Ιούνκερ μίλησε για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για τα θέματα αυτά. Το ερώτημά μου είναι τι θα γίνει με τις πληρωμές που εκκρεμούν από τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ώστε να πιστεύω ότι θα μπορέσουν να καλυφθούν αυτές οι πληρωμές τα επόμενα χρόνια και δεν υπάρχουν ε, λόγοι να πιστεύουμε ότι θα μειωθούν όλα αυτά τα πράγματα αυτόματα τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο να αλλάξει αυτή την πολιτική που έχει να συνάπτει συνέχεια πιστώσεις υποχρεώσεων, υποχρεώσεις ενώ περικόπτει τις πιστώσεις πληρωμών. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες προσπάθειες και να το εγγράψουμε αυτό και στην ενδιάμεση αναθεώρηση, γιατί αλλιώς θα παραμείνει σε επίπεδο μεγαλεπίβολων σχεδίων η περιφερειακή πολιτική, αλλά δεν θα επιτύχει τίποτα σε επίπεδο εφαρμογής. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κομισιόν μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν πράγματι τη δυνατότητα σε συνεργασία να διευρύνουν ακόμα περισσότερο την συνεργασία των περιφερειών και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα με τι παραμεθόριες περιοχές. Ελπίζω λοιπόν κύριε Επίτροπε ότι και στο νέο σας, στα νέα σας καθήκοντα θα μπορέσετε να διευρύνετε ακόμα περισσότερο την συνεργασία μεταξύ παρομεθωρίων περιοχών και βλέποντας ποια είναι η κατάσταση σε πολλές από τις χώρες που είναι όμορες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες διαπεριφερειακής συνεργασίας έθεν και εκείθεν των συνόρων. Ελπίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν τις περιφέρειες που βρίσκονται στα σύνορα των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόν, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επιτρόπο κύριο για τον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζεται τη περιφερειακή πολιτική τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπάρχει μια ομάδα κρατών μελών, ε, του φίλου τη συνοχή, όπω του λέμε. Δεν είναι όμω δυστυχώ όλα τα κράτη-μέλη φίλοι τη συνοχή και κάνατε εσεί καταπληκτική δουλειά προασπιζόμενο στην πολιτική συνοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σα ευχαριστήσω για τη βοήθεια που δώσατε τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ουαλία. Ξέρω ότι ε, κάνατε επισκέψεις, ε, είδατε διάφορα σχέδια, προγράμματα, ξέρετε ότι στην Ουαλία έχει μεγάλη σημασία να έχουμε αυτά τα κονδύλια συνοχή και βέβαια μπορείτε να μα επισκεφτείτε όποτε θέλετε και στο μέλλον. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τι συμφωνίε εταιρική σχέση. Θα πρέπει να υπάρχουν αυτέ οι συμφωνίε και θα πρέπει και οι τοπικέ αρχέ, οι περιφερειακέ αρχέ να συμμετέχουν. Πιστεύετε όμως ότι σε τέτοια χάρη τον κώδικα συμπεριφοράς, ε, λειτουργήσε σωστά ή τελικά δεν εφαρμόζεται καλά από τα κράτη-μέλη και μένουν στα λόγια. Και κάτι άλλο, πώς μπορούν οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές ε, με μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω να συμμετέχουν περισσότερο στους κανονισμούς ε, και στα κοινά σχέδια δράση λοιπά, θεσμικές επενδύσεις, όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει, είναι νέοι μηχανισμοί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θα ήθελα την άποψή σα, λοιπόν. Τα κράτη-μέλη εκμεταλλεύονται τις νέες αυτές δυνατότητε, αυτού του νέου μηχανισμού ή μένουν στα λόγια μόνο. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπεθ. Ε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε, για τη δουλειά σας. Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση το τελευταίο... Ε, πρέπει... Δυστυχώς όχι, δεν πρέπει, διότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η ανισότητα, η ανεργία, η φτώχεια, υπάρχουν διαφορές. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά που γίνεται. Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν ειδικά σε κάποιες χώρες ε, δημιουργούν δυσκολίε, η οικονομική ανάπτυξη δεν υπάρχει και παράλληλα, επειδή δεν υπάρχει, δημιουργούνται ε, θύλακες ε, φτώχειας, ανισότητας. Πρέπει να σκεφτεί επ' αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων μου δημιουργεί πολλές ελπίδες που ανακοίνωσε ο, η Επιτροπή και ο πρόεδρο Γιούνκερ. Αλλά πρέπει να πω ότι δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί η Ευρώπη ε, ξεχνάει τους, τις βασικές αρχέ αρχές και δημιουργεί ανισότητες. Ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα και ως Ήπειρο έχουμε τεράστιο, κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε ε, μια ολόκληρη γενιά, τους νέους, τους λιγότερο ε, έτοιμους, ε, να τους αφήσουμε πίσω μας Κομισιόν, θεωρείτε ότι αυτές οι πολιτικές λιτότητας, ε, κοινωνικών περικοπών, δεν έχουν ε, επίπτωση στην αύξηση της ανισότητας στην Ευρώπη, ειδικά ε, σε προγράμματα, που είναι υποδια... προγράμματα διάσωσης, σε χώρες που είναι προγράμματα διάσωσης. Ε, αυτές οι πολιτικές μπορεί να είναι συμβατές με την ολοκλήρωση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη μείωση της στόχιας και της ανισότητας. Ευχαριστώ. κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Επίτροπε, είμαι νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά από το 1998 μέχρι και σήμερα ε, δραστηριοποιήθηκα έντονα στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, διατέλεσα δήμαρχος, ήμουν και υπουργός της Σλοβανική Κυβέρνηση και θέλω να σας συγχαρώ για το έργο σας και για το τι έχετε επιτύχει στο ε, πεδίο της πολιτικής συνοχής. Θα ήθελα να πω ότι η πολιτική συνοχή σε διάφορες πτυχές, υποδομές, ανάπτυξη τουρισμού, ευρυζωνικότητα για τις περιφέρειες, αξιοποίηση των πηγών ενέργειας κτλ. Όλα αυτά νομίζω ότι πράγματι τόνωσαν την ανάπτυξη στα κράτη-μέλη, ιδίως εν καιρό κρίσης. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ε, μερίδιο της χρηματοδότησης που δόθηκε στη Σλοβενία. Βέβαια, έχω επιφυλάξει προς το ότι το 1 τρίτο ε, των πόρων δεν τα έχουμε ακόμη, δεν το έχουμε αξιοποιήσει και υπάρχουν ε, και συμφωνίες συνδέσεις που εκκρεμούν, δεν έχουν υπογραφεί ακόμη. Πρέπει μέχρι το τέλος της να έχουμε εξελίξεις θετικές και θα ήθελα να καλέσω και όλα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Και έτσι θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε με τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2011. Πρέπει να στηρίξουμε τις υποδομές, ε, η πολιτική συνοχή από την άλλη. Θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει υποδομές, τη διασύνδεση μερικών ε, απομακρυσμένων περιοχών, τη σύνδεση διαξηράς θαλάσσης κτλ. Και πρέπει και τα κράτη-μέλη, Σλοβενία και Κροατία, να συνδεθούν πιο αποτελεσματικό. Ο κ. Μποστινάρου έχει τώρα το λόγο. Κύριε Επίτροπε, πάρα πολλά ωραία λόγια ακούστηκαν προς το πρόσωπό σας ε, δικαιολογημένα και θα προσθέσω και εγώ τις δικές μου ευχαριστίες ε, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε την τελευταία πεντέτια. Χάρη σε εσά και στην ομάδα σας κύριε, ο Νικόλας Μάρτιν, Πίτερ Μπέρκοβιτς, είχαμε μια πραγματικά γνήσια σύμπραξη. Καλάξαμε το πρόσωπο της πολιτικής συνοχής και εγώ θέλω να φέρω μόνο τρία σημαντικά στοιχεία. Σκονόμηση ενέργειας Υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή στη σχέση μας με τη Ρωσία, αλλά είναι άκρος επίκαιρο το θέμα. Επίσης, η διευκόλυνση συνάντας στην Ευρώπη, το Connecting Europe Facility, είναι κάτι σημαντικό. Και τρίτον, θεσμική ικανότητα, διοικητική ικανότητα, πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την απαιτούμενη προσοχή και τα απαιτούμενα μέσα. Το ερώτημα μου όμως είναι το εξής. Σήμερα που εγκαταλείπεται αυτή τη θέση. Πώς αξιολογείται την ικανότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν αυτό το μέσο, αυτή τη διευκόλυνση συνέντα στην Ευρώπη πριν τα τέλη του Δεκεμβρίου 2016 και από 1η Ιανουαρίου 2017. Και βέβαια να σας ευχαριστήσω γιατί στηρίξατε και την πρόταση των Ρωμανικών Αρχών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης προσέγγισης στο σχέδιο του Δέλτα του Δούναβη. Τόσο σημαντικό για μας όχι μόνο για τη χώρα μου, αλλά και για την Ευρώπη εν γέννη. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Μπρέσου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Και από μένα για τη δουλειά που κάνατε. Και καλή επιτυχία στα νέα σας αξιώματα. Σίγουρα θα σας δούμε και εκεί. Μία ερώτηση μια και εσείς μας αφήνετε έτσι... Κάνετε μια αποτίμηση για τη δουλειά που κάνατε όλη αυτή τη διάρκεια. Έχουμε τώρα πολλές μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Πώς συντονίζονται αυτές με την πολιτική συνοχής. Γιατί από τη μία έχουμε ένα προγραμματισμό και από την άλλη ένα διαφορετικό προγραμματισμό. Από την εμπειρία σας, τι έχετε να πείτε αφιερώνουμε καθόλου πόρους για, για, τον προγραμματισμό των, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή είμαστε ακόμα σε επίπεδο λόγων και εξαγγελιών. Στην πραγματικότητα δεν συνδέονται ακόμα με την συνοχή. Ο κύριος Βαλκάθερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παναγία. Κύριε Επίτροπε, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τη συνοχή, για εταιρικές σχέσεις, ε, για σπατάλες κτλ. Είμαι καινούριο όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, αλλά όπως ξέρετε κι εσείς και οι συνάδελφοι και ο Επίτροπος ε, Χαν, επί 19 μέλη, ε, χρόνια ήμουνα μέλος της Επιτροπής των, Περιφερειών Γίνω και πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών. Ο κύριος Χάν έκανε μία αναφορά σε αυτά που είπε η κυρία Μπρέσο και σε άλλους. Ε, σας ευχαριστώ που είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Θέλω να πω στον Επίτροπο Χάν και στους υπόλοιπους συναδέλφους ότι δεν ήταν καθόλου δύσκολο να συνεργαστούμε με τον Επίτροπο Χάν τα τελευταία χρόνια. Ήταν εύκολη η συνεργασία. Γιατί? Γιατί ακούσαμε με άμεσο τρόπο πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όταν έχουμε απέναντί μας έναν επίτροπο με ευαισθησίες, με διάθεση για συμβιβασμούς κτλ. Ένας συνάδελφος από την Κροατία μίλησε για τις πλημμύρες στην Κροατία. Ε, θυμάμαι κάτι που συνέβη ε, στη δική μου περιοχή, στη Μούρθια, στην Ισπανία, στην Νόρκα. Μάλιστα υπάρχει και ένας Ισπανός ποιητής με αυτό το όνομα. Στην τρίτη πόλη της Μούρθια το 2011 έγινε ένας καταστροφικός σεισμός με πολλούς θανάτους και κατέστρεψε και μια ιστορική περιοχή, ε, πολλά μνημεία της περιοχής αυτής, δυστυχώς. Πρέπει να πω ότι αμέσως κινητοποιήθηκαν διάφοροι πόροι, διάφορες βοήθειες για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό της πόλης αυτής που ήταν σε απελπισία. Ο Επίτροπος Χάν έθεσε και κονδύλια στη διάθεση των κατοίκων από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Όχι μόνο έκανε αυτό, όχι δηλαδή έδωσε μια πολιτική απάντηση, αλλά ε, είχε και μια ανθρώπινη παρουσία. Αυτά γιατί σας μίλαγα προηγουμένως για ευαισθησία και για διάθεση να δει τα πράγματα από κοντά. Πήγε στη Μούρφια ο Επίτροπος, πήγε στην, ε, στην πόλη του Λόρκα και μας έδωσε ελπίδα ε, με τη ζεστασιά του κτλ. Ε, ήταν εκεί ως άνθρωπος. Δεν θέλω να μιλήσω για, ούτε για βιομηχανική μετατροπή, ούτε για συνοχή. Θέλω απλώς, γι' αυτό πήρα το λόγο, να σας ευχαριστήσω, να αναγνωρίσω τη θαυμάσια δουλειά που κάνατε και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο, φαντάζομαι και, και εγώ όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, στα νέα σας καθήκοντα. Ε, σε αυτό το νέο αξίωμα, ευρωπαϊκό και αυτό, που είναι μπροστά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εγώ θα ξαναγυρίσω όταν ξαναγυρίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτι το οποίο με ζητά, μου ζητάνε να εξηγήσω και εγώ ίδιος δεν γνωρίζω και εγώ ίδιος νιώθω σύγχυση μερικές φορές γιατί ήμουν στον επιχειρηματικό κόσμο πρωτού έρθω εδώ και όχι στον κυβερνητικό χώρο. Όταν λέτε ότι υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού, μιλάμε για 23,4 δισεκατομμύρια τα οποία εκκρεμούν αλλά συνεχίζουν τα σχέδια, η εφαρμογή τους. Αν το κάνατε αυτό στον επιχειρηματικό κόσμο, θα τρώγατε μια κλωτσιά ή τουλάχιστον θα σας αποχαιρετούσαν. Σε αυτό το σενάριο όμως που είμαστε λέτε θέλουμε περισσότερα λεφτά, μα όταν αποφασίζεται ένας ο προϋπολογισμός υπάρχει μια σύνδεση στις νοητικές διαδικασίες μεταξύ των χρημάτων που είναι διαθέσιμα και το τι θέλετε, πόσα θέλετε να δαπανίσετε ή αυτό γίνεται, γίνεται τελείως ανεξάρτητα η διαδικασία και μόνο μετά πάτε να τα συμβιβάσετε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για όλα τα ερωτήματα. Κύριε Επίτροπε, λιγότερο από 10 λεπτά έχετε να απαντήσετε όλα αυτά τα συνολικά και πολυπληθή ερωτήματα. Αλλά έχουμε άλλη μία παρέμβαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το μόνο που ήθελα να ρωτήσω ήταν ένα σύντομο ερώτημα προς τον κύριο Επίτροπο. Κύριε Επίτροπε, ποια είναι η αποψή σας σε ό,τι αφορά την ε, μέθοδο της ανάπτυξης που ξεκινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς βλέπετε το ρόλο αυτής της μεθόδου στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, γιατί η μεν επιγνώση του γεγονότος ότι η Κομισιόν προώθησε στο παρελθόν αυτή την μέθοδο. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν για μια μορφή ανάπτυξης η οποία έλκεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο στο μέλλον και κατά τα άλλα σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο μελλοντικό σας έργο. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Όχι, όχι, δεν θέλετε να αρρωστεί και άλλα ερωτήματα. Νησάφι πλέον. Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις σας κύριε Επίτροπε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά σε ό,τι αφορά. Την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, το πολύ. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στον κανονισμό, στους κανονισμούς μας και φαντάζεστε ότι η εφαρμογή της ιδέας αυτής δεν είναι το ίδιο τα, δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κρατη Ξαρτάται βέβαια από τις θεσμικές ε, δομές σε κάθε κράτος. Βέβαια έχει ξεπεράσει τις δικές μου προσδοκίες η χρήση του. Ο Λιφαντεμ Μπράντε, εκ των τέως προέδρων της Επιτροπής των Περιφερειών, ήταν ένας από τους ε, σκαπανείς της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης Περιμένουμε μια έκθεσή του τις επόμενες εβδομάδες. Του ζήτησα να εκπονήσει αυτή την έκθεση και να είναι έτοιμη αυτή μέχρι τα τέλη της χρονιάς, το αργότερο, για να διατηρηθεί αυτή η ορμή, ο καλός ρυθμός και έτσι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αλλά και να προκαταλάβουμε ενδεχομένω τα αποτελέσματα για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού βέβαια θα πρέπει να χτίσουμε πάνω στο ότι έχει γίνει μέχρι τώρα. Όπως είπα δεν ε, έκαναν τα ίδια όλα τα κράτη-μέλη, αλλά πιστεύω ότι έχουν σεβαστεί ή έχουν αρχίσει να, να σέβονται αυτή την ιδέα. Σε ό,τι αφορά αυτά τα 300 δις, φυσικά τα διαρθρωτικά ταμεία θα διαδραματίσουν ένα ρόλο μεταξύ πολλών άλλων γιατί υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βέβαια από την πλευρά της ε, που μπορεί να παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση. Αλλά θέλω να επαναλάβω και κάτι που είπε και στην ε, εισαγωγική μου ομιλία. Μπορώ πραγματικά να ζητήσω και να παρακαλέσω σχεδόν τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν περισσότερο τις δυνατότητες που τους δίνουν τα χρηματοδοτικά μέσα για να υπάρχει η απαιτούμενη μόχλευση Και αν χρειαστεί, ίσω δεν αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια να έχουμε ένα ποσό άνω των 300 δι. Ό,τι αφορά το διορθωτικό προπολογισμό, είπαν κάποιοι ε, συνάδελφοί σα ορισμένα πράγματα. Είναι πολύ πλοκο το θέμα γενικά με την κατάρτιση του προπολογισμού. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Εμείς έχουμε τηρήσει όλους τους κανονισμούς και τα σχετικά. Υπάρχει όμως ένα όλο και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων. Το οποίο προκαλείται και από το ότι στις νέες μεσονομικές προοπτικές εισάγεται αυτό η αρχή του νησιν 3 και για την οροφή, την αιτήσια οροφή των πληρωμών. Επομένως, δεν είναι τόσο, θα έλεγα, θέμα χρηστής μεσονομικής διαχείρισης, όσο ανάγκης ε, να τηρούμε τις πολιτικές δεσμεύσεις και συμφωνίες. Άπαξ και συμφωνείται λοιπόν ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, από εκεί και πέρα οι αιτήσεις και προπολογισμοί αντιστοιχούν σε μια κατανομή του πολιετούς αυτού προγραμματισμού και ο προπολογισμό αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τι συμφωνίε που ελήφθησαν για όλη την διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών. Και βέβαια ε, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Και αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο τα διαφορετικά ταμεία, θα επηρεάσει όλε τι γραμμέ, όλα τα κονδύλια του προπολογισμού, γεωργία, ορίζοντα 2020, εξωτερικέ σχέσει τα πάντα. Δεν περιορίζονται τα προβλήματα στο κόστος άλλων πολιτικών και α, ε, τούμπαλιν, λίγο πολύ θα επηρεάσει με διαφορετικές διαβαθμίσεις σε απόλυτα νούμερα όλες τις πολιτικές. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόβλημα ειδικό που αφορά μόνο τη δική μας πολιτική, αλλά αφορά όλες τις πολιτικές. Όταν εκταμιεύονται ε, χρήματα και επιστρέφονται στα κράτη-μέλη. Και θέλω να περάσουμε και ένα μήνυμα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες έχουμε έναν προπολογισμό. Από αυτόν τον προπολογισμό, περίπου το 6% μόνο το 6% το χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όχι μόνο οι κομισιόν, μισθή, δικαστήριο, ελεκτρικό κτλ. Τα πάγια έξοδα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν ξεπερνάνε το 6% του ευρωπαϊκού περιπολογισμού και πάνω από 94% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για δραστηριότητες στα κράτη-μέλη. Το 94% είναι ένα μικρό κομμάτι για δραστηριότητες εκτός Ένωσης, αλλά το 94% και παραπάνω επαναλαμβάνω για δράση, ενέργειες, για project, για έργα. Και όλοι μαζί πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτή την αναλογία. Για μια πώς να την πω, κερδοσκοπική επιχείρηση, μια εταιρεία. Μπορεί να πει μια εταιρεία ότι έχει τέτοια αναλογία παγίων και λειτουργικών δαπανών και να υπερηφανευτεί για αυτήν. Γι' αυτό λοιπόν δεν ζητούμε πρόσθετους πόρους για τους πολίτες μας ή για τις υποδομές. Εμείς ζητάμε απλά τα χρήματα αυτά για να αποζημιωθούν, να τους επιστραφούν δηλαδή ε, οι δαπάνες αυτών που έχουν προχρηματοδοτήσει, προκαταβάλει τα ποσά. Και κυρίως μιλάμε για ιδιώτες ή ε, για εταιρείε, ε, τελικούς δικαιούχους που περιμένουν, περιμένουν τα χρήματα. Και υπάρχει κίνδυνος πτώχευσης, χρεοκοπίας για ορισμένους λόγω ακριβώ αυτών των καθυστερήσεων. Γι' αυτό και ε, θέλω την κατανόησή σας. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε χρηστή κατάρτιση προπολογισμού κάθε χρόνο. Ε, βέβαια είμαι και λίγο συναισθηματικά φορτισμένο για αυτά τα θέματα, αλλά πρέπει να το προσέχουμε το θέμα του προπολογισμού. Για τον κύριο Βον, για την Ουαλία, την συμφωνητέρικη σχέση. Α, δεν είναι εδώ. Έφυγε. Τέλος πάντων. Αυτό το πω για τους υπόλοιπους. Τα μέσα που έχουμε προτείνει εφαρμόζονται διαφορετικά ανάλογα με τις δομές, τις ιδέες των κρατών μελών. Γενικά όμως ε, είμαστε ικανοποιημένοι για τον κύριο Μπλάνκο Λόπεθ. Είναι δύσκολο να πει κανείς τι θα είχε γίνει αν δεν υπήρχαν τα τα μία. Υπάρχει ταμεία. Υπάρχει μια ένδειξη βέβαια. Πριν την κρίση, τα διαθροτικά ταμεία αντιστοιχούσαν στο 7% του συνόλου των δημοσίων επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και τους καθόλου φορείς μιλάω. Μετά την κρίση, και ελπίζω πλέον να μπορούμε να μιλάμε για το μετά την κρίση, τέλο πάντων, σήμερα, για να το πω αλλιώ, τα διαθετικά ταμεία έχουν φτάσει στο 20% των ε, δημοσίων επενδύσεων στην Ευρώπη. Τριπλασιάστηκε δηλαδή το ποσοστό σε σχέση με την εποχή πρώτης κρίσης. Η σημασία και ο ρόλος των εθνωτικών ταμείων. Είναι σημαντικό γιατί ε, αποζημιώνει για την έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων. Μιλάμε για 600.000 ε, θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν και ίσως μετά το τέλος περίοδο να μπορούμε να μιλάμε και για 1,4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Σίγουρα δεν έχουν αντισταθμίσει εντελώ οι απώλειε και οι χαμένε θέσει εργασία, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά στο μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης για μια ακόμη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε και πάλι απευθυνόμαι στα κράτη-μέλη. Μιλάμε τόσο πολύ για αυτή την πρωτοβουλία για την νεολαία. Έχουμε δώσει 6 δισεκατομμύρια. Τα εκταμιεύσαμε γρήγορα σχετικά θα έλεγα, αλλά να σας πω κάτι. Μόνο το 25% Αυτόν των 6 δισεκατομμύρων μέχρι στιγμής έχουν δοθεί για, την, για τις διάφορους διαγωνισμούς. Δίνονται οι πόροι, αλλά μέχρι στιγμής μόνο το 1 τέταρτο αυτών των κονδυλίων, το 25% έχει χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό ζητώ να το χρησιμοποιήσουν τα κρατημέρια αυτά ποσά με διαγωνισμούς, με δημόσιες προμήθειες κτλ. Γενικά τώρα. Ευφύης εξειδίκευση, διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί να εκπαιδεύουμε κόσμο να τους προσθέτουμε δεξιότητες αν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας που να μπορούν να διεκδικήσουν. Είναι η πρόκληση αυτή και θα δείτε τις επόμενες χρονιές, είμαι βέβαιος, τα αποτελέσματα των πολιτικών μας γιατί θα αυξηθούν ε, οι δυνατότητες. Έρχομαι στο φίλο μου τον κύριο Ποστινάρου. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας και ευγενικά λόγια, όπως και τους άλλους βέβαια συναδέλφους σας. Είμαι γενικά αισιόδοξο. Πιστεύω ότι οι διοικήσεις βελτιώνονται όλο και περισσότερο. Φυσικά και θα επενδύσουμε στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, νομίζω πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι καλά δεν τα λέω, ναι, για την περαιτέρω Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης είναι υπαρθών 11 προτεραιότητα. Είμαι πεισμένος και αισιόδοξο ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τις ε, διοικήσεις μας για να συμμορφωθούμε προς όλες τις απαιτήσει. Μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Μια πρώτη αξιολόγηση δείχνει ότι πράγματι τα κράτη-μέλη έχουν ε, από εκ των προτέρων λάβει υπόψη τους τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και έχουν ε, αφήσει κατά μέρο ποσά για αυτές. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια και για την έρευνα. Δεν κατάλαβα βέβαια ακριβώ πώ το εννοούσατε, αλλά εγώ θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι στι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ θα είναι στενή η συνεργασία μεταξύ αυτών που εργάζονται στην έρευνα και αυτών που απασχολούνται στα διαφορετικά ταμεία και στην Ευρώπη αλλά και στις χώρες μέλη. Έχουμε να διδαχθούμε πολλά από τον άλλο. Υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες, διαφορετικές εμπειρίες. Όμως, παρόλα αυτά, είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε κοινό έδαφος για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και ιδίως για να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια ανεπάρκεια και δυναμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι άλλη από την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ έρευνας, ε, έκβασης της έρευνας και επιχειρηματικών ευκαιριών. Εδώ λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο, αλλά είμαι αισιόδοξο. Ότι τα μέσα, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και οι πόροι οικονομικοί θα επαρκέσουν. Αλλά αν είμαστε ευφύς και πρέπει να πω και πεισματάριδες, ισχυρογνώμονες. Να εφαρμόσουμε δηλαδή ε, στην πράξη τις κοινέ μας ιδέες και να υλοποιήσουμε τα συμπεφωνημένα. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την πάρα πολύ επικοδομητική, τουλάχιστον για εμένα, πενταετία και όπως φαντάζεστε θα χύσω παραπάνω από ένα δάκρυ όταν θα σας εγκαταλείψω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής, να σας ευχαριστήσω για την προσωπική σας συνεισφορά, για την υπεράσπιση και εφαρμογή των πολιτικών, των πολιτικών μας. Ε, σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στα μελλοντικά σας καθήκοντα. Τώρα, κλείνω το δημόσιο τμήμα της συνεδρίασής μας και περνάμε στο κομμάτι κεκλεισμένων των θυρών. Ε, όποιος δεν είναι συντονιστής, όποιος δεν δικαιούται να είναι παρόν, παρακαλώ να βγει από την αίθουσα. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο.